Dear colleagues, if you want to take your places, we can... Αν θέλετε να ξεκινήσουμε, θα έρθουν και οι υπόλοιποι σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξέρετε κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι προσκεκλημένοι, χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Γραφείου Εισαγγελίας, του ΕΠΠΟ και του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας, Eurojust. Έχουμε τον κύριο Λίζερμαν εδώ που εκπρόσωπη την ε, Ολλανδία. Έχουμε την κυρία Γκρέσλε, την Επιτροπή Ελεγχτών Προϋπολογισμών. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας η κυρία Σιλίφεν Κάουφμαν, ε, ενεργό μέλος Επιτροπής μας, ο κύριος Νίκολας Φράνσεν από την Ολλανδική Προεδρία Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για τον Τερνισμό EPPO και η κυρία Αλεξάνδρα Ζουρ Σρότερ διευθύνουσα σε θέματα ποινικού δικαίου από τη Γενική Διεθνή Δικαιοσύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίση να αναφέρω πω έχουμε και μια ομάδα Αυστριακών δημοσιογράφων μαζί μα. Καλώ ήρθατε. Ο Χάιντ Σπέκερ, ο συνάδελφο, καλό συνάδελφο Χάιντ Σπέκερ, του έχει προσκαλέσει εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ελπίζω να σας ε, κινήσει το ενδιαφέρον αυτή η συνεδρία, ίσως να μην είναι τόσο συναρπαστικά αυτά που θα ακούσετε σήμερα σχέση με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα σας, αλλά Ελπίζω να σας ενδιαφέρουν παρόλα αυτά. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η θέσπιση της EPPO, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, εισαγγελία είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη και ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της απάτης και της, ε, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξού και η σχετική ακρόαση σήμερα από την πρόταση του Ιούλιο του 2013 σχετική με τον Κορισμό, το Κοινοβούλιο ζητάει από, τον, από το Συμβούλιο να διαφυλάξει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική νομιμότητα, ενημερώνοντα τακτικά, ζητώντα τακτικά τη γνώμη του Κοινοβουλίου και λαμβάνοντα τι ε, γνώμη τη θέση του υπόψη. Είναι ζήτημα ε, μεγάλη σημασία εν ώψη τη έγκριση του Ευρωπαϊκού κανονισμό για την ΕΠΠΟ. Έχουμε εν προκειμένου υιοθετήσει το Μάρτιο του 2014 και το Μάρτιο του 2015 αντίστοιχα δύο ψηφίσματα που υπογραμμίζουν ιδιαίτερα την ανάγκη για μια πλήρω ανεξάρτητη αρχή ΕΠΠΟ για την προστασία των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και μια σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΠΠΟ και των Εθνικών Εισαγγελικών Αρχών. Θα ήθελα προκειμένου να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες σχετικέ με ε, αδικήματα απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την οδηγία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και των απατών, τη λεγόμενη οδηγία PIF. Η έγκριση της οδηγίας αυτής αποτελεί και προϋπόθεση για την συνένεση στην έγκριση του κανονισμού. Πολύ εξημών γνωρίζεται ασφαλώς ε, πως οι συνομιλίες ε, σε επίπεδο Συμβουλίου συνεχίζονται και έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλευρά του Συμβουλίου. Θα έχουμε έναν Ευρωπαίο ε, εισαγγελέα από κάθε κράτος μέλος σε μόνιμες συνθέσεις στην ΕΠΠΟ και θα οργανώνονται έτσι οι υπηρεσίες σε σχέση με τις εθνικές ε, εισαγγελικές υπηρεσίες σε πρώτη φάση. Λοιπόν και στο πρώτο τμήμα της συνεδρίας θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για τη λειτουργία της EPPO, την αντιμετώπιση των αδικημάτων της οδηγίας PIF. Ε, τα ε, επιτεύγματα της Eurojust είναι νομίζω σημείων μεγάλη επιτυχία, σηματοδοτούν μεγάλη επιτυχία, έχουν να κάνουν και με το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και κυρίως τις δικονομικές ε, διασφαλιστικές δικλείδες για τη διεξαγωγή της ποινική δίκης και αυτό βέβαια πάντα αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα, ύψιστη προτεραιότητα για μας εδώ στην Επιτροπή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, η σχέση μεταξύ της PPO, της Eurojust, της Όλαφ επίσης, θα έλεγα, ε, έχουν μεγάλη σημασία και θα πρέπει να υπάρξει σαφή διαφοροποίηση και διάκριση των ρόλων των τριών αυτών υπηρεσιών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών αυτών για να είναι αποτελεσματική καταπολέμηση των αδικημάτων ε, που περιγράφει η οδηγία PF. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι τη συναντησή μα για το Κοινοβούλιο. Ο κανονισμό οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζει συνοχή στην καταπολέμηση και την δίωξη των εγκλημάτων και των ε, αυτούργων του σε σχέση με τις ποινικές αυτές διαδικασίες στο δικαίωμα για ε, δικαστική αποκατάσταση θα πρέπει πάντοτε να είναι στο στόχαστρο του κάθε του ΕΠΠΟ Έτσι, κάθε απόφαση που θα λαμβάνει η ΕΠΠΟ θα πρέπει να υπάγεται σε μια δικαστική αξιολόγηση πριν να προχωρήσει η υπόθεση στα δικαστήρια ε, δικαστήρια κράτους μέλους ή Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αντίστοιχα, πράγμα το οποίο πάντα είναι περίπλοκη υπόθεση και θα συζητηθεί και αυτό μεταξύ των εμπειρογνωμόνων μας, τελική μας συζήτηση, το τελικό τμήμα της συζήτησης. Καλωσορίζω λοιπόν πρώτα εκ μέρους της Προεδρίας, η οποία εκπροσωπείται σε ολόκληρη την ακρόαση, όπως είπα, τον κύριο Άιζερμαν. Αναπληρωτή διευθυντή, Γενικό Διευθυντή για την ε, επιβολή του νόμου, εκπρόσωπο της Ολλανδικής Προεδρίας σε θέματα ποινικά και έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Thank you very much. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω τη σύντομη εισαγωγική μου παρέμβαση στην ακρόση, εκφράζοντας τη, τη συγνώμη μου μάλλον, γιατί ο Υπουργό Βαντεστούρ, που είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Συντερικών και Δικαιοσύνης, δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να παραστεί σε αυτή την εκδήλωση, λόγω κατεπηγουσών ανηλυμένων υποχρεώσεων. Τώρα στο θέμα μας. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Προεδρία της Ολλανδίας έκανε ό,τι μπορούσε για να πετύχει αυτή πρόοδο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, βασιζόμενη βέβαια, επί του έργου προηγουμένων Προεδριών. Και αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ με κάθε μετριόφροσυνη νομίζω ότι έχουμε πετύχει κάποια πράγματα. Ξεκινώντας, ήδη μπορούσαμε να πλησιάσουμε συμφωνία όσον αφορά τις γενικές διατάξεις περί στελέχωσης και κόστους εν ώψη του Συμβουλίου Εσωτερικών και δικαιοσύνη στις 11 Μαρτίου και συζητήθηκε η πολιτική όσον αφορά την έννοια της επιχειρησιακής δαπάνης, της ενίας της επιχειρησιακής δαπάνης. Μετά το Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης συζητήσαμε εκτενώς την όλη διαχείριση και το σύστημα διαχειρήσεων υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων που έπρεπε να αφιγραμμιστούν με το πρόσφατο πακέτο για την προστασία των δεδομένων, καθώς και εναλλακτικέ όσον αφορά τη δίωξη. Ένα θέμα που αναφέρεται ως συναλλαγές επισήμως το θέμα ως προστασίας των δεδομένων είναι μάλλον περίπλοκο. Δοθήσεις της θέσεως κάποιων κρατών μελών. Αυτά ανησυχούν για τη δυνατότητα που υπάρχει μεταξύ, συγκρούσεως μεταξύ των κανόνων προστασίας δεδομένων για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διατάξεις όσον αφορά τη δική τους νομοθεσία για το ποινικό δίκαιο. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε αλλά το θέμα ίσως να απαιτήσει περαιτέρω συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο πριν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα σε αυτή τη φάση. Μετά το Συμβούλιο της 9ης Ιουνίου Εσωτερικών και δικαιοσύνη θα παρουσιάσουμε ό,τι θα είναι έτοιμο να παρουσιαστεί στους ε, υπουργούς σαν μια μερική γενική προσέγγιση τότε πλέον η επόμενη, η Σλοβακική Προεδρία θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει τις ε, διαπραγματεύσεις. Όμως ε, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας κάτι. Είναι περιπλοκότατο το ζήτημα. Υπάρχουν αποκλίνωσες απόψεις και υπάρχουν και μεγάλα συμφέροντα από πλευράς κατών μελών. Το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετάσχουν. Δεν σας εκπλήσει ότι το Ολλανδικό μας Κοινοβούλιο παρακολουθεί εκ του το θέμα και έχει ακόμα επικρίνει, έχει μια διστακτική θέση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία. Θα ήθελα να πω ότι έχει ολοκληρωθεί η εργασία του Συμβουλίου. Το πνεύμα ήταν ένα καλό θετικό πνεύμα συνεργασία. Στόχο ήταν να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα επιτρέπει στα περισσότερα κράτη-μέλη θέλουν και μπορούν να συμμετάσχουν. Αυτό πιστεύει η Προεδρία θα είναι κρίσιμη σημασία και για αποτελεσματικότητα και για αξιοπιστία τη μελλοντική αυτή, Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία. και αυτό έχει μεγάλη σημασία ούτω ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική ε, αντιμετώπιση της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, σε αυτό το τομέα, πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Σας διαβεβαιώνω ότι όλες οι αντιπροσωπείς στο Συμβούλιο μελέτησαν προσεκτικά τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι συστάσεις αυτού ε, συζητήθηκαν εις βάθος της διαπραγματεύσης. Πιστεύω ότι τώρα έχετε μια καλή εικόνα των εξελίξεων από όταν ξεκίνησε η Προεδρία μας και θα ήθελα να κλείσω με μια σύντομη δήλωση λέγοντας ότι προσβλέπω σε μια ενδιαφέρουσα ακρόαση σήμερα το απόγευμα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα Πάμε στο πρώτο θέμα, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής που θα αντιμετωπίζει την απάτη και τα εγκλήματα αποτελεσματικά. Πρώτο πάνελ. Έχω τη χαρά να καλωσορίσω τη κυρία Ingeborg Γκρέσλερ που είναι ε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, και, Κοντ και έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω ιδιαίτερως να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την συμπερίληψη στην ημέρα διάταξη αυτού του σημαντικού θέμα, διότι νομίζω ότι θα μα οδηγήσει στην επιτυχία το να συζητούμε διαρκώ τα αισθήματα αυτά και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Ολλανδική Προεδρία. Ιδιαίτερα εκτιμούμε τι προσπάθειε σα και του ε, κόπου σα. χωρί ο οποίο δεν γινόταν τίποτα. Χαίρομαι βεβαίω όταν λέτε ότι ότι θέλετε να ολοκληρώσετε τις ε, διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας είναι πολύ σημαντικό αυτό και θετική είδηση για όλους μας γιατί περιμένουμε χρόνια τώρα να δούμε την ολοκλήρωση αυτής της υπόθεσης ε, και κάθε εξάμεινο περιμένουμε να δούμε τα βήματα, τα μικρά βήματα που θα προωθήσουν προς τα μπρος την υπόθεση αυτή. ευχαριστούμε λοιπόν και θέλω να σας διαβεβαιώσω για την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Του προπολογισμού. Έχουμε λοιπόν ε, με την κυρία Λόπε Αγγιλάρ και την κυρία Τσίπρη επίσης ε, μοιράσει αυτή την υπόθεση μεταξύ μας. Συνεργαζόμαστε στενά οι δύο επιτροπές, διότι θέλουμε ιδιαίτερως να, να δώσουμε τη διασύνδεση μεταξύ του κανονισμού υπό και, του, και της οδηγίας PIF για την ποινική δίωξη ε, αδικημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ρυθμίζονται οι καθήλυνα αρμοδιότητε της Ευρωπαϊκής ε, Η διασύνδεση βρίσκεται στο άρθρο 17 του σχεδίου κειμένου του Συμβουλίου για τον κανονισμό ΕΠΟ, εκφράζεται εκεί, όπου περιγράφεται η διασύνδεση μεταξύ των δύο ε, διαδικασιών αυτών, νομοθετικών αυτών διαδικασιών. Το θέμα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, θεωρούμε ότι η ΠΙΦ έχει πολύ μεγαλύτερη, ε, προσφέρει μεγαλύτερε δυνατότητε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί αυτή η διάσταση ιδιαίτερω στη διαδικασία. Όπω λέμε λοιπόν, όπω λέει και ο συγητή, είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία ΠΙΦ και είναι ε, σημαντική η διάκριση. Δεν πρέπει να υπάρξουν ε, ως προς τις καθήλυνα αρμοδιότητες διαφοροποίησης στον κανονισμό ΕΠΟ και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τα κείμενα όπως έχουν κατευθεί μέχρι στιγμής, ε, αν και θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση της Αγγελικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ πιο ορθολογική σε σχέση με αυτό το οποίο προέκυψε ύστερα από επίπονε διαπραγματεύσει επίπεδο Συμβουλίου. Οι συντρέψει λοιπόν αρμοδιότητε τη ΕΠΟ και των Εθνικών Αρχών, για τι οποίε δίνει μεγάλη σημασία το Συμβούλιο, ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικέ, γιατί έτσι μπορούμε να ε, πούμε ότι δεν θα έχουν το δικαίωμα τα κράτη-μέλη να επαναπαύονται και να σταυρώνουν τα χέρια όταν διαπιστώνουν τα χρήματα στα, τα, τα οποία έχουν ε, ε, χαθεί λόγω καταχρήσεων, είναι μόνο ευρωπαϊκά χρήματα. Πρέπει λοιπόν να δραστηριοποιηθούμε για την καταπολέμηση αυτών των καταχρήσεων. Σε σχέση με τον περίπλοκο χαρακτήρα των διατάξεων και των αρμοδιοτήτων που ορίζει ο κανονισμός ΕΠΟΚ με τις συμπληρωματικέ διατάξεις 17, 18, 20 και 22α τα σχετικά άρθρα, ε, ιδιαίτερα ε, προβληματικό βλέπουμε το κείμενο της ε, διάταξης του άρθρου 23β το οποίο λέει ότι δεν έχει αρμοδιότητα η ΕΠΟ όταν υπάρχει άλλο θύμα πλήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ύψος ε, ποσού ισοδύναμο ή υψηλότερο από τη ζημία που έχουν υποστεί ε, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν θα έχει αρμοδιότητα σε περίπτωση χρηματοδότηση κατά 50% ή περισσότερο με ευρωπαϊκά κονδύλια, σε περίπτωση εμπορίου γιατί η χαμένη τελωνιακή δασμή θα είναι πολύ χαμηλότερη από τους εθνικούς ε, φόρους, ε, ο φόρος προσθέμενης αξίας γιατί έστω και αν έχει κάποια βασική αρμοδιότητα για τον φόρο προσθέμενης αξίας η ΕΠΟ θα είναι πολύ μεγαλύτερο το μερίδιο που θα πηγαίνει στον εθνικό προπολογισμό από αυτόν και βεβαίως δεν είναι δυνατόν ε, ο εθνικός σύνδεσμος όπως ονομάζεται να λειτουργήσει αποτελεσματικά, δηλαδή οι Ευρωπαίοι εισαγγελεί να, έχουν, ε, να παρακολουθήσουν την ίδια υπόθεση και στο κράτος μέλος και γι' αυτό θα έπρεπε και για λόγους ε, επιμερισμού της, ε, του ε, φόρτου να έχει τη δυνατότητα ένας, εθνικός, ένας ευρωπαϊκός εισαγγελέας να στήσει από τον ε, Chief Prosecutor την ανάθεση σε κάποιον άλλο από τους αδέλφους του της παρακολούθησης μιας υπόθεσης σε σχέση με την οδηγία PIF Προσπαθούμε να προωθήσουμε την οδηγία. Έχουμε μέχρι τώρα καταφέρει αρκετά καλά αποτελέσματα. Σε ένα σημείο έχουμε ζητήματα μόνο, το φόρο προσθέμενης αξίας, όπου τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται να καταλήψουν συμφωνία, αλλά νομίζουμε ότι για λόγους και συστηματικούς πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Έχουμε κοινού ορισμούς λοιπόν, τι είναι το οικονομικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι είναι οι καταχρήσεις και οι απάτες σε σχέση με επιδοτήσεις και διαγωνισμούς, νομοποίηση παράνομων εσόδων, κατάχρηση κονδυλίων κοινοτικών, ενεργή και παθητική διαφθορά, τι είναι οι υπάλληλοι, τι είναι οι εντολοδόχοι. Δεύτερο στοιχείο της οδηγίας είναι ο προσδορισμός κοινών των ε, συνθήκων και ε, προδιαγραφών για τις ε, κυρώσεις και τις ελάχιστες τιμές. Μεγάλη σημασία βέβαια θα έχει η αντιμετώπιση του ζητήματος του φόρου προσθεμένης αξίας, όπως είπα και νωρίτερα, ε, και είπα ότι θα πρέπει να, και θέλω να υπογραμμίσω ότι χρειάζεται να καλύπτεται το φόρο προσθεμένης αξίας σε περίπτωση όπου αφορά η διαφθορά τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη ή ζημία τουλάχιστον 100.000 ευρώ ή ε, Ευρωπαίο υπάλληλο ή μέλη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Μέχρι τώρα αρνείται κατηγορηματικά το Συμβούλιο να συμπεριλάβει το θέμα του φόρου προσθεμένη αξία στις συζητήσεις του. Θα δούμε αργότερα Τώρα σε σχέση με τα opt-out την αυτοεξαίρεση δηλαδή και το ΠΙΦ, το σύστημα της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση διαφθοράς θα κρυθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτά, μεγάλο πρόβλημα ε, σε σχέση με τις ε, θέσεις μας ως Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει να κάνει με το ότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης αυτών των συνθήκων. Έχουμε την αλλαγή της νομικής βάσης από το 325 στο άρθρο 83 της Συνθήκης Ατλητουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πηγαίνει στην δικαστική συνεργασία αντί της ε, ε, πρώτης νομικής βάσης η οποία θα σήμαινε υποχρεωτική συμμετοχή όλων των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν έχουν τη δυνατότητα κάποια κράτη-μέλη να αυτοεξαιρεθούν. Αναμένεται ότι τουλάχιστον τρία θα αυτοεξαιρεθούν και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολλέ διαφορετικέ δομέ κατά πολέμη διαφθορά ε, από ε, ορισμένα κράτη. Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Αναμένουμε βέβαια τη νέα οδηγία ΠΥΦ ε, για 25 κράτη-μέλη. Η παλαιά σύμβαση ΠΥΦ του 1995 ε, θα εξακολουθήσει να ισχύει όμως για τα τρία κράτη-μέλη που έχουν το opt-out. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος με, με τον κανονισμό EPPO να μην συμμετέχουν ορισμένα κράτη, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει ακόμα μεγαλύτερο κατακαιρματισμό και συνέπειες. Ο κατακαιρματισμός των θεσμών επίση των υπηρεσιών και των οργάνων ε, που ε, καθίσταται ακόμη πιο ορατός και προφανή σε σχέση με την Όλαφ και εδώ νομίζω ότι τίθενται διάφορα ερωτήματα στα οποία πρέπει να δοθούν από απαντήσεις. Δηλαδή η Όλαφ στο μέλλον πώς μπορεί να οργανώνεται εσωτερικά δεδομένου ότι στο, στην επικρα... Τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένα κράτη-μέλη, για διαφορετικά κράτη-μέλη, θα υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες θα λειτουργούν παράλληλα. Και πώς θα μπορεί σε περίπτωση περισυνοριακών υποθέσεων η Όλαφ, Φερρυπίν, η με ένα βασίλειο, κάποιο άλλο κράτος που έχει το opt-out της ε, σύμβασης PIF του 1995 ως νομική βάση ή το ε, Βέλγιο ή και το Βέλγιο Φερρυπίν με τη νέα οδηγία PIF. Πώς θα αντιμετωπίσετε τις περιπτώσεις ε, η Όλαφ, εάν οργανωθεί έπω ορισμένα λόγη σε όλα, πάντα θα υπάρχουν πάντα ε, κάποια προβλήματα σε σχέση με τι συνοριακέ υποθέσει και βεβαίω και το προσωπικό θα επηρεαστεί από αυτό και η στελέχωση των υπηρεσιών. Όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν και θα ήθελα κλείνοντας ε, με ένα θετικό μήνυμα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΠΟ και της Όλαφ. Έχουμε το άρθρο 57 α, το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Όλαφ που θα πρέπει να διατηρηθεί για να μπορεί να αναλαμβάνει ε, διερεύνηση υποθέσεων ε, ανεξαρτήτως του αν ε, το επιθυμεί και η ΕΠΟ, να μπορεί η Όλαφ να αναλαμβάνει κατά πρωτοβουλία δική της έρευνας ανεξαρτήτως του αν το δέχεται ή αν μπορεί να το ακολουθήσει και η ΕΠΟ. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε υποστήριξη της, ΕΠΟ, της Όλαφ βεβαίως όταν έχει ανάγκη από αυτήν η ΕΠΟ. Ε, θα ήθελα επίσης με όλες τις δυσκολίες που έχω υπογραμμίσει να μην ε, αφήσω αρνητικές ε, εικόνες και εντυπώσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν καλές λύσεις που μπορούν να προχωρήσουν και ελπίζουμε ότι θα έχουμε στο τέλος με τη συνεργασία με το Συμβούλιο ένα καλό κείμενο πριν φτάσουμε στη τελευταία στιγμή γιατί εκεί θα χρειαστεί να αρχίσουμε από το ε, μηδεν Το τρίγωνο αυτό, ΕΠΟ, Eurojust και Όλαφ ε, θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται με ιδιαίτερε δυσκολίε. Πρόκειται για ένα τρίγωνο συνεργασία το οποίο θα πρέπει να δώσει θετικά αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε πόρους ε, που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με τρόπο οικονομικό και δεν μπορούμε να ε, κατασπαταλούμε τους πόρους μας. Ε, για να είμαι αισιόδοξη λοιπόν κλείνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ελπίζω σύντομα να έχουμε μια συμφωνία και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού έχει κάθε καλή διάθεση να συνεργαστεί. Βέβαια θα κρατηθούν τα πάντα από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια από τα ζητήματα τα οποία θέσατε. Φαντάζομαι θα μας τα απαντήσει η Σιλβή η Φων Κάφμαν, επόμενη ομιλήτρια, η οποία θα μιλήσει εκ μέρους του κ. Λόπεθ Αγγιλάρ, που ήταν ο συνεισηγητής της ΛΥΜΠΕ για την οδηγία ΠΥΦ. Η Σιλβή Ιβών συμμετείχε ενεργότατα σε όλη αυτή τη σχετική δίκηση του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, σου δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Κλόντα. Κύριε Πρόεδρε, όντω ο κύριο Λόπε Αγγελάρη, ηγητή για την οδηγία ΠΙΦ, δεν μπόρεσε να είναι σήμερα παρόν μαζί μα και έτσι στο σημείο αυτό αναλαμβάνω εγώ να πω δύο λόγια σε σχέση με τη θέση μας ε, και τη θέση των ομάδων στην υπόθεση αυτή. Κάθε χρόνο χάνονται έσοδα από το ΦΠΑ, από ε, τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και από τα κράτη-μέλη. Και εδώ ιδιαίτερη σημασία έχει να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα. Όπως είπε και η κυρία Γκρέσλε, υπάρχει ε, διάκριτική συμφωνία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης του 1995. Ωστόσο υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση διαφθοράς, ε, του ιζωμοποίηση παράνομων εσόδων, των απατών στην ευρωπαϊκή και, αντίστοιχα διαφορετικέ ποινικέ διαδικασίε. Υπάρχουν σημεία λοιπόν αδυναμία ε, ω προ ε, τα συστήματα ελέγχων, ε, η ανταλλαγή πληροφοριών πέραν των συνόρων μεταξύ κρατών, η ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών είναι ο, ο αυτών των φαινομένων. Η κοινωνία λοιπόν απαιτεί την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των ε, περιπτώσεων διαφοράς ε, και δεν υπάρχει κατανόηση γιατί πρέπει να μείνει στο ε, από τις ιστορίες αυτός ο αγώνας για την καταπολέμηση της, Ευρωπαϊ... της διαφθοράς σε σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο πολίτης ε, περιμένει δίκαια ολογημένα να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του η Ευρωπαϊκή Ένωση και να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα. Ο τριμερής διάλογος συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια. Πρόκειται για διαπραγματεύσεις οι οποίες ε, νομίζω ότι αξίζει να εκτεθούν σε, σε σχέση με ορισμένα σημαντικά στην ΧΙΑ. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με, ευρωπαϊκούς κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε σχέση με τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα που πρέπει να εναρμονιστούν, να προχωρήσουν παράλληλα. Εμείς, κατά κύριο λόγο, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, βλέπουμε ε, αδύρυτο δεσμό μεταξύ της ΠΙΦ και της, και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό όμως προϋποθέτει ταυτόχρονα και την εξασφάλιση των όρων της αρμοδιότητάς της ε, Ευρωπαϊκής Αγγελίας πρέπει να, πρέπει να δοθούν λοιπόν οι ορισμοί ώστε να είναι ξεκάθαρο γιατί πράγμα έχει την καθέλη αρμοδιότητα αυτή η εισαγγελία και θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω πως, έχουμε να κάνουμε, πως εδώ η έγκριση της οδηγίας ΠΥΦ αποτελεί προϋπόθεση για υποστήριξη από πλευράς μας ε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έγκρισή της. Δεύτερον, η ομάδα Σοσιαλιστών Δημοκρατών ε, ε, υπογραμμίζει ιδιαίτερο την σημασία του φόρου προσθεμένης αξίας ως πηγής εσόδων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το ανέφερε και η κυρία Γκρέσλε, έχει κεντρική σημασία ανέκαθεν και πάντα και έχει να κάνει όχι μόνο με την καταπολέμηση τη απάτη σε σχέση με τα, ευρωπαϊκά, με τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την προστασία των ιδίων πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση Τάρικο στις 8 Σεπτεμβρίου ε, του 2015 αποφάσισε πως η άμεση συνεργασία με, ε, σχέση με την ίσπραξη ε, του ΦΠΑ έχει να κάνει με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία ΠΥΦ λοιπόν καλύπτει κατά εμάς την, τα θέματα του φόρου προσθεμένης αξίας και αντίστοιχα υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για την δίωξη τέτοιων εγκλημάτων και με βάση αυτή την απόφαση Τάρικο, διαρωτώ με πως είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη ακόμη να μην έχουν δείξει την αντίστοιχη ευελιξία σε σχέση με τα μέτρα αυτά. Ένα άλλο σημαντικό σημείο σε σχέση με την οδηγία PIF είναι οι ελάχιστες ποινές για συγκεκριμένα αδικήματα. Πρέπει να προσοριστούν αυτές Τη ε, τις προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο με την εκθεσή του υποστήριξε τις προτάσεις αυτές. Ελάχιστες λοιπόν ποινές, οι οποίες υφίστανται και σε άλλα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματι στην οδηγία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου εις βάρος ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε εδώ με ένα πάρα πολύ σημαντικό και κεντρική σημασία ζήτημα, στο οποίο χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι τα κύρια, τα τρία ε, κεντρικά σημεία ε, για μας ε, αυτής της οδηγίας. Έτσι μπορεί να οργανωθεί η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και κυρίως αυτού της, της ε, λεγόμενης κυκλικής απάτη σε σχέση με το ΦΠΑ. Πρόκειται για τον αγώνα του κυρίου Λόπες Αγγιλάρ, ο οποίος θα συνεχιστεί βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σύρβια. Θα ακούσουμε την Ολλανδική Προεδρία, τον κύριο Νίκολα Σασάνσιν που είναι Πρόεδρο τη ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Έχετε το λόγο για ένα δεκάλεπτο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την πρόσκληση που απευθύνατε προς την Ελληνική Προεδρία να παραστεί στην ακρόαση. Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής. Στο ρόλο μου έχω σαν πρόεδρο για 47 ημέρε της ομάδας εργασίας για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εξ αρχής ότι η Ολλανδική Προεδρία εξέτασε αρκετά ζητήματα από την πρώτη πρώτου, αλλά όχι με τα συγκεκριμένα άρθρα που αφορούν την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής. Είναι κάτι που είχε συζητηθεί πριν ξεκινήσει η δική μας Προεδρία, του του το παρόν κείμενο για τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα το βρείτε σε ένα έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε στο τέλος της Λουξεμβουργικής Προεδρίας το 151-00 κάθετος 15 και βασίζεται επί της ιδέας κοινή αρμοδιότητας μεταξύ του EPPO και των εθνικών διοκτικών αρχών, εισαγγελικών αρχών. Βασιζόμαστε επί πρακτικών λόγων για κάτι τέτοιο. Θα ήταν πολύ δυσχερές και χρονοβόρο αν κάθε υπόθεση που εξετάζει ένα τοπικό εισαγγελέα πρέπει να διαβιβάζεται στον Ευρωπαϊκό εισαγγελέα. Κυρίω αν ο, ο ντόπιο εισαγγελέα μπορεί ε, να, ολοκληρώσει την... να διεκπαιρεώσει την υπόθεση γρήγορα και αποτελεσματικά μόνο του. Θα ήταν πολύ δύσκολο από την αρχή μια έρευνα να γνωρίζει κανεί αν μια υπόθεση ε, ανοίξει αρμοδιότητα του ΠΙΦ ή αφορά εθνική απάτη ή όχι. Εάν ο χαρακτήρας πιφ της υποθέσεως αποδειχθεί σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, δεν έχει νόημα να αφήσουμε τον εθνικό εισαγγελέα να εγκαταλείψει την υπόθεση και να τη διαβιβάσει στο ΕΠΠΟ. Το παράδειγμα των αδικημάτων των, ε, ε, θα έπρεπε να αναφέρεται. Σε κάποια κάτι μέλη ίσως να υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις που αφορούν λαθρεμπόριο μικρών ποσοτήτων ενοπνεύματος κάθε χρόνο. Λαθρεμπόριο βότκας, από τα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας ε, θεωρείται ότι είναι με τέτοια υπόθεση. Κάθε τέτοια υπόθεση ενδεχομένως αποτελεί ένα δίκημα πιφ. Θεωρείται ότι δεν είναι αποτελεσματικό να μεταφερθούν, να διαβαστούν στο ΕΠΠΟ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή υποθέσεις και κάποια άλλα τελωνιακά δικήματα δεν ε, ανήκουν σε μια κατηγορία μακροχρονίων ποινικών ε, διαδικασιών. Άρα όλα αυτά τα επιχειρήματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται η κοινή αντιμετώπιση από εθνικές αρχές και η ΠΠΟ. Όμως η Ευρωπαϊκή Αγγελική Αρχή, το ΕΠΠΟ, θα έχει προτεραιότητα όσον αφορά ε, την δίωξη υποθέσεων ΠΙΦ. Δηλαδή θα ενημερώνεται το ΕΠΠΟ για όλες τις υποθέσεις ΠΙΦ που διαπιστώνουν τα κράτη-μέλη και τότε θα αποφασίσει να τις ζητήσει να διαβαστούν από τις εθνικές εισαγγελικές αρχές ή όχι προφανώς. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Υπηρεσίας πιο συγκεκριμένα σε υποθέσεις που αφορούν τις βλάβες και ζημίες προς τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κάτω από 10.000 ευρώ αυτά τα δικήματα θα παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο καταρχήν εκτός αν υπάρχουν συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι ύποπτοι είναι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η οι υποπτοι ειναι αξιωματουχοι τη Ευρωπαϊκή δεν πληροπατορισμονή, ουδή. η ευρωπαικη εισαγγελια θα έχει πάντα το δικαίωμα να αναλαμβάνει όλε τι σημαντικέ υποθέσει πιφ. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονεί Η Προεδρία είναι πεπισμένη ότι αυτή η λύση εγγυάται ισορροπημένο και αποτελεσματικό σύστημα όσον αφορά τι αρμοδιοτητε όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει το γενικό έλεγχο και την εποπτεία των περισσότερων υποθέσεων πιφ. Όμως ταυτόχρονα μπορεί να εστιάζεται επί των σοβαροτέρων υποθέσεων. Ούτως τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν να αντιμετωπίσουν υποθέσεις πιφ με διαφορετικό τρόπο αν ο τρόπος αυτός είναι αποτελεσματικότερος εφαρμόζοντας διοικητικές, επιβάλλοντας διοικητικές κυρώσεις Φερρυπίν. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του ΕΠΠΟ σε ρατσιόνε ματέριε, Πράγματι, όπως και ήδη ανέφερε η κυρία Γκρέσλε, το άθρο 17 καθορίζει ότι η οδηγία πιφ όταν θα έχει εγκριθεί και εφαρμοστεί θα καθορίζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Αγγελική Αρχή θα είναι αρμόδια σε σχέση με ποινικά δικήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Απάτε Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και απάτε που έχουν διαπραχθεί στα πλαίσια μια εγκληματική οργανώσεω σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αλληλένδετα δικήματα καλύπτονται και από αυτή τη διάταξη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή έχει αρμοδιότητα για αυτά τα δικήματα, θα το δείτε στο άρθρο 20, παράγραφος 3, εκτός εάν η μέγιστη κύρωση για το δίκημα πιφ είναι λιγότερο σοβαρή από τη μέγιστη ποινή για την στενά, αλληλένδετη, άρρηκτα συνδεδεμένη, συνδεδεμένο αδίκημα. Η κύρωση είναι ίση εκτός εάν το άλλο αδίκημα είναι βασικό για τη διάπραξη του αδικήματος πιφ. Ή όπως είπε η κυρία Γκρές, η ζημιά στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν ξεπερνά τη ζημία προς άλλο θύμα που είναι κάτι που αφορά το θέμα της συμπερίληψης του ΦΠΑ ή όχι. Τέλος, επί του σημείου αυτού είναι σημαντικότατο να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ΕΠΠΟ και των εθνικών αρχών, οι εθνικές αρχές θα έχουν τον τελικό λόγο. Όσον αφορά το κρίσιμο θέμα για τις απάτες το θέμα του ΦΠΑ, αν οι απάτες ΦΠΑ συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία ΠΙΦ ή όχι, εν ίδια απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας ε, Γκρέσλε, αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Όμως η Ολλανδική Προεδρία είχε τρεις συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο όσον αφορά αυτό το θέμα για να βρούμε μια λύση και θα παρουσιάσουμε τα πορίσματα των συνεδριάσεων στο Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στις 9 Ιουνίου. Αυτό ούτως ώστε να υπάρξει συμφωνία επιβάσεως διαπραγματεύσεων για συζητήσεις μάλλον διαπραγματεύσεων το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εδώ να προσέξουμε κάτι. Πρέπει να πω ότι κατέστησα σαφές ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές αντιδράσεις από πλευράς αρκετών κρατών μελών όσον αφορά τη συμπερίληψη των απατών στον τομέα του ΦΠΑ. Να υπογραμμίσω ότι τα κράτη-μέλη εκείνα επουδενή δεν διαφωνούν όσον αφορά την ανάγκη να καταπολεμηθεί απάτη όσον αφορά το ΦΠΑ και μάλιστα με ζήλο, αλλά φρονούν ότι υπάρχουν αποτελεσματικότεροι τρόποι καταπολέμησης απάτης αυτής. Πολύ συχνά αυτό ισχύει στη μορφή συνδυασμού διοικητικής αντιμετώπισης με αντιμετώπιση μέσω του ποινικού δικαίου. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας και σας κύριε Πρόεδρε για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα πάμε στην τελική παρουσίαση του πρώτου τμήματος Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Αλεξάνδρα Ντύρ Σρόντερ, Διευθύντρια για τα θέματα ποινικού δικαίου στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Έχετε το λόγο μέχρι ένα δεκάλεπτο. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, να σας καλησπερίσω. τη βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ που δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τελευταία το λόγο. Συνήθω είμαστε οι πρώτοι που παίρνουμε το λόγο, αλλά έχουμε τώρα το πλεονέκτημα, αν θέλετε, κάπω και να συνοψίσουμε την όλη συζήτηση. Και να πω ότι ήδη ορισμένα από αυτά που ήθελα να αναφέρω έχουν ήδη υποθεί. Οπότε θα ήθελα απλά να αναφέρω νέε ιδέε. Εστιάζω καταρχά ε, στην ουσιαστική αρμοδιότητα του, Ευρωπαϊκή της για την οδηγία ΠΥΦ. Έχω προετοιμάσει τρει ε, διαφάνειε ε, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και την παρουσίασή μου, αλλά πρώτα απ' όλα μία επενθύμηση. Το ακούσαμε από τους ομιλητές του πάνελ ε, αν υπάρχει αποκλειστική συντρέχουσα αρμοδιότητα. Θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχική της πρόταση ξεκινούσε από ε, αποκλειστική αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ίσως να ε, είχαμε δει τα πράγματα λίγο άσπρο-μαύρο ό,τι αφορά το αποκλειστικό ή όχι και καταλαβαίνω και τις ανησυχίες της κυρίας Γκρέσλε ότι η πρόταση δεν διευκολύνει τα πράγματα ε, όσοι έχει τώρα. Και το έχουμε συζητήσει διαμακρών με το Συμβούλιο και είναι γνωστά τα επιχειρηματά του. Τα έχουμε λάβει υπόψη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ουσιαστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφή. Θα πρέπει να εκπηγάζει απευθεία από την οδηγία PIF. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος αδικημάτων στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διότι πρόκειται για μια δυναμική αναφορά, δυναμική μνήμα. Και θέλω να πω ότι επειδή είχαμε συζητήσεις και με τα κράτη-μέλη για το κατά πόσον θα ήταν ίσως καλύτερο να συμπεριληφθεί αυτό στον κανονισμό της Αγγελίας ή η προσέγγιση της Κομισιόν που ήταν να μπει ε, στην οδηγία ΠΙΦ, μήπως αυτό παραβιάζει τη συνθήκη διότι ο κανονισμός ΕΠΟ, ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απαιτεί ομοφωνία καθότι κανονισμός. Εμείς όμως δεν θεωρούμε ότι υπάρχει νομικό κόλλημα για την χρήση αυτής της τεχνικής, ώστε να έχουμε μια οδηγία που θα ορίζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είπε η κυρία Κάφμαν ότι χρειάζεται ευρωπαϊκό πλαίσιο για δικήματα στο πλαίσιο τη οδηγία ΠΛΙΦ. Και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απολύτω μαζί σα, κυρία Κάφμαν. Αυτό είναι και ο στόχο τη ε, Κομισιόν ε, με την πρόταση αυτή τη οδηγία ΠΙΦ πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο για να προστατευτούν καλύτερα τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ εντάσσονται κάποιε πτυχέ που θα ήθελα να συντομία να αναφέρω. Καταρχά, Εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε ένα μέσο ποινικού δικαίου που είναι πάνω από 20 ετών, η οδηγία δηλαδή του 95, 21 ετών λοιπόν, άρα απερχιωμένο και σε ό,τι αφορά την νομική τεχνική έχουμε το, ε, την ομολογία πλέον, έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τα ποινικά δικήματα και θα πρέπει να δούμε και πώς τα δικήματα ή αν θέλετε αξιόπινη συμπεριφορά έχει εξελιχθεί μετά την οδηγία PIF. Κάτι άλλο σημαντικό. Τι είναι public official, αυτή η έννοια πρέπει να οριστεί. Γιατί τα δικήματα PIF πολλές φορές δεν πράττονται από ε, δημόσιους αξιωματούχους, γιατί μιλάμε για δημόσιο χρήμα. Οι κανόνες για τις κυρώσεις σημαντικό κομμάτι έχουν να δραματίσουν στο ποινικό δίκαιο. Να σας πω, ε, παρενθέσει, ότι στην πρότασή μας είχαμε για πρώτη φορά προτείνει ε, την εισαγωγή των ελάχιστων κυρώσεων, αλλά μάλλον ήταν πρόημο ε, κάτι τέτοιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και για το Συμβούλιο, δεν μπορούσαν να το δεχθούν. Για μας αυτό είναι κρίμα, γιατί θεωρούμε ότι θα είχε αποτρεπτικό αποτέλεσμα, αποτρεπτική ισχύ. Κάτι τελευταίο, η οδηγία αυτή περιλαμβάνει και τους κανόνες για την παραγραφή και για τις ε, ε, περιόδους ε, ισχύσεις προθεσμίες. Δεν θέλουμε να καινοτομήσουμε έτσι και μόνο. Απλά πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές αυτά τα αδικήματα έχουν μια συγκεκριμένη έτσι πολύ ιδιαίτερη σχέση με το χρόνο και γι' αυτό πρέπει κάπως να τα ρυθμίσουμε. Τώρα, για τα ποινικά δικήματα ορισμός είναι λίγο πολύ αυτό στη σύμβαση ΣΠΙΦΑ για την απάτη, παραδείγματος χάρη, και έχουμε και μια νέα έννοια ε, fraudulent activity, δούλια δραστηριότητα, απατηλή δραστηριότητα. Ε, ε, δωροδοκία, το embezzlement, άλλα δικήματα όπως διαφθορή, διαφθορά, corruption, money laundering, ξέπλυμα χρήματος ο χρηματισμός. Όλα αυτά είναι σημαντικά και πρέπει να τα λέμε υπόψη. Να δούμε και τα έσοδα με τι δαπάνε. Θέλουμε να έχουμε ένα πλήρε πλαίσιο. Συγγνώμη, embezzlement, υπεξαίρεση. Και επίση ε, να αναφέρω κάποια από αυτά που ανέφεραν προλαλήσαντες Μπορεί να τα έχουν ξαναπεί, αλλά πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι η απάτη ΦΠΑ πρέπει να ενταχθεί ε, στα περί των χρηματοοικονομικών συμφερόντων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη θέση της Κομισιόν πράγματι έχουμε καλά επιχειρήματα που ευσταθούν και νομικά αλλά και είναι και από πολιτικές πλευράς ε, στέρεα. Θεωρούμε δηλαδή ότι η απάτη ΦΠΑ πρέπει να συμπεριληφθεί. Από ηθικής πλευράς. Θεωρούμε ότι είναι λογικό να ενταχθούν τα σχετικά δικήματα στην οδηγία. Τώρα, θα σα θέσω ένα ερώτημα και δεν θα, μπορώ, δεν θα ήθελα να δώσω ε, μια τελική απάντηση σήμερα. Πώ όμω ε, θα περιλάβουμε αυτέ τι υποθέσει ε, απάτη ΦΥΠΕΑ, θα τι περιλάβουμε έτσι όσο έχουν στην οδηγία ή ίσω σκοπιμότερο θα ήταν να περιοριστεί η οδηγία σε σοβαρέ ε, υποθέσεις απάτη ΦΠΑ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή σήμερα, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το εξετάσουμε αφού θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει ε, στο πλαίσιο μέρο διαλόγου και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε ένα καλό σημείο αναφορά. Αν, σοβαρά θέλουμε, ε, να, αν θέλουμε να δούμε το θέμα αυτό σοβαρά, θα πρέπει να βρούμε και το κατάλληλο benchmark για να καθορίσουμε το κατόφλι. Και στην τελευταία διαφάνεια πάντα για την απάτη ΦΠΑ, πώς μπορούν να συνάδουν ε, η οδηγία ΑΠΙΦ και ε, δεν μπορώ να σας δώσω απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα σήμερα. Θα θέσω και εγώ ε, τα δικά μου ερωτήματα προς εσάς. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι αν θα πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ πεδία εφαρμογή τη οδηγία για, για τι απάτες ΦΠΑ και τι αρμοδιότητε ε, του ΕΠΟ τη Ευρωπαϊκή Αγγελία ε, σε μια ιδανική περίπτωση και την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να ήταν ταυτόσιμο το πεδίο εφαρμογή δηλαδή, αλλά υπάρχουν περιθώρια συζήτηση μεταξύ των ε, συνομοθετών για το θέμα αυτό. Αυτό όμως που δεν θεωρούμε ότι είναι η ορθή προσέγγιση είναι να χρησιμοποιηθεί ήδη η έννοια τη το, το διασυνοριακό ε, στην οδιαπίφη, Διότι μιλάμε για απλικά μέσα, μιλάμε για την ουσιαστική αρμοδιότητα, material competence. Και νομίζω ότι αυτό το υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ε, στην ελληνική δικονομία. Δεύτερο ερώτημα λοιπόν είναι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει αρμοδιότητα για ορισμένα μόνο ε, αδικήματα που έχουν να με το ΦΠΑ και που σχετίζονται με κάποια κράτη-μέλη, πέραν του ενός ενδεχομένω. σίγουρα να ζητούμε και εμείς ε, ε, λογικές, συμβιβα... Ε, λογικές συμβαστικές προτάσεις που όμως θα διατηρούν την ουσία της πρότασης της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά και τον κανονισμό ΕΠΟ και σε ό,τι αφορά την οδηγία ΠΙΦ, πάντα σε θέματα απάτης ΦΠΑ. Νομίζω ότι ήμουν εντός του χρονικού ορίου. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, να πράγματι σας και ξέρετε γιατί, ξέρετε γιατί μου το είπατε, γιατί είμαι πάντα αυστηρός μέσα με τον χρόνο. Δεν το κάνω επίτηδες. Ε, ευχαριστώ πάντως όλους και όλες που ήσασταν πολύ ε, συνοπτικοί. Έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις. Το χαρτί μπροστά μου όμως προς το παρόν είναι λευκό. Δεν έχει κανείς ζητήσει το λόγο. Περίεργο αυτό. Τι έγινε, σας κάναμε μάγια. Συνήθως πολλοί είναι αυτοί που θέλουν το λόγο. Πάντω πρέπει να πω πάρα πολύ ευσύνοπτες, πάρα πολύ πλήρηση παρουσιάσεις. Αχ, Μπάρμπαρα, μπράβο, σε ευχαριστώ που σήκωσες το χέρι σου. Μόνο για σένα, Κλοντ, μόνο για σένα. Θέλω να ρωτήσω. Είναι το εξής. Μήπως έχουμε υποχώρηση ε, μια εκένωση, αν θέλετε, ενός ε, πολύ φιλόδοξου σχεδίου του άρθρου 86 των συνθήκων, κυρίως παράγραφος 4 που συνέστηνε την αύξηση των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα διεθνή εγκλήματα, τα υπερεθνικά εγκλήματα. Μία υποχώρηση και δυστυχώς το Ευρωκοινοβούλιο έχει ελάχιστη εξουσία να το αντιμετωπίσει. Μόνο εκφράζει απόψεις. Διερωτώ με. Τι, ποια είναι η ακριβής μας λειτουργία. Γιατί μιλώ για υπαναχώρηση και επιδείνωση. Όσο περνάει ο χρόνος, η πρόταση για την ευρωπαϊκή η εισαγγελία φαίνεται να αντιγράφει κάπως το, τη μοίρα του Eurojust. Να μην έχουμε επιχειρησιακό οργανισμό, αλλά ένα οργανισμό που ελέγχει και συντονίζει τις ε, δράσεις των εθνικών εισαγγελικών αρχών. Ίσως κάνω λάθος, αλλά θα ήθελα πάνω σε αυτό να γνωρίζω ε, ποια είναι η υποψή σας. Το επιβεβαιώνετε αυτό ή το διαψεύδετε. Δηλαδή, Είμαστε ενώπιον της δημιουργίας ενός σώματος με εκπροσώπους που θα καθορίζονται από τα κράτη με έναν κατάλογο αρμοδιοτήτων ανεξαρτήτων ε, στο ελάχιστο δυνατό και με μια τάση να να επιστρέφουν οι αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη, όλο και περισσότερες. Δηλαδή, αρμοδιότητες που αρχικά θέλαμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Σαγκυρική Αρχή να επιστρέφουν στα κράτη-μέλη. Θα είναι ένα κολέγιο, ένα σώμα, όπου τελικά οι ελεγχόμενοι γίνονται ελεγκτές. Θα σταματήσω εδώ και θα ρωτήσω αν όσον αφορά την ανάλυση μου για αυτή την υποχώρηση έναντι των μεγάλων προσδοκιών που είχαμε και του εγχειρήματο που ξεκινήσαμε, κάνω λάθος για την εικόνα αυτή που έχω σχηματίσει. Ευχαριστώ. Μπρίγκετ Σίπλ. Ευχαριστώ. Κλοντ. Θα ήθελα να συνεχίσω σε ένα άλλο σημείο και θα αναφερθώ στο σημείο που αναφέρε ο πρόσωπος του Συμβουλίου ότι ελπίζει όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν. Εγώ θα έλεγα αντίθετα ότι με ένα τέτοιο νομοθέτημα και κυρίως το κόστος που θα συνεπάγεται αυτό πρέπει να συμμετάσχουν όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κράτη. Και θα διαφοροποιηθώ και σε σχέση με την κυρία Κρέσλε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχει αλλάξει η Επιτροπή Λίμπε τη νομική βάση αλλά ότι υπάρχει η δυνατότητα της αυτοεξαίρεσης. Απλώς και μόνο αυτό. Αυτό πρέπει να απαγορευτεί. Ε, δεν νομίζω ότι κατά τα άλλα θα έχει αντίρρηση κυρία Γκρέσλε. Τώρα στο εάν θα συμμετάσχουν όλα τα κράτη-μέλη. Ήδη εξετέθη το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Εάν δηλαδή θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι υπάρχει λόγος ανάληψης δραστηριότητας, τι είδους μέτρα έχει ή θα πρέπει να στήσει από τον Εθνικό Εισαγγελέα, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη να κάνετε την έρευνα και εκείνο μπορεί να αρνηθεί, οπότε δεν θα γίνεται η έρευνα. Ή αλλιώς θα χρειάζονται νέα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η διασπάθηση χρήματο. Και βέβαια εδώ, όπω συμβαίνει κάθε φορά που αναμειγνύονται προ τα κράτη-μέλη, το κριτήριο θα πρέπει να είναι το ποιο θα αποφασίσει και ποιο θα είναι το κριτήριο στο οποίο θα καταλήξει μια υπόθεση διαφιλονικούμενη για λόγους ε, αρμοδιότητας ε, η οποία καταλήξει στα δικαστήρια λόγω αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού ε, Εισαγγελικού Γραφείου για να μην έχουμε ένα forum shopping εν τέλει. Ευχαριστώ Μπίρκετ. Μπάρμπαρα Ματέρα, εισηγήτρια εκ μέρους του, της Επιτροπής μας για την ΕΠΠΟ. Και εγώ θέλω προς τον κύριο Φράντσα να απευθύνω την ερώτησή μου. Θα ρωτήσω κατά πόσο το Συμβούλιο σε τεχνικό επίπεδο έλαβε υπόψη την υπόθεση να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Συγγελία πριν εγκριθεί η οδηγία PIF. Αν αυτό συμβεί, θα δημιουργηθεί μεταβατική κατάσταση εν αναμονή της οριστικής εγκρίσεως της οδηγίας PIF. Ευχαριστώ. Και στο τρίτο τμήμα των συζητήσεων θα καθοδηγείτε τις συζητήσεις. Λοιπόν, ας απαντήσετε με τη σειρά στις ερωτήσεις, αλλά παρακαλώ λάβετε υπόψη και τόσα είπαν άλλοι συνάδελφοι. Σίγουρα θα ακούσατε κάτι το οποίο θέλετε να θίξετε και να αναλύσετε. Θα ακολουθήσετε μια σειρά που θα σας ε, δώσω. Η κυρία Γκρέσλες ξεκινήσει λοιπόν. Α, όχι. Ναι. Ναι, ναι. Θέλω κι εγώ μια ερώτηση μάλιστα. Για την κυρία Σουρέτερ. Στην αλληλεγγύη της νομικής βάσης. Είχε συζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ενδεχομένο να προσφύγει κατά του Δικαστηρίου και του Κοινοβουλίου για το θέμα της νομικής βάσης. Νομίζω ότι δεν είναι κακή ιδέα. Είναι γνωστό ότι σε ορισμένα θέματα επιμένω αρκετά. Και γιατί, γιατί ε, σε μεγάλο βαθμό η επιλογή της νομικής βάσης είναι υπεύθυνη για το χάος στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, το νομικό. Ε, η αναποτελεσματική αυτή οργάνωση βεβαίως δεν θα επιτρέψει την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δεσπάθησης ευρωπαϊκού χρήματος από τους ε, ελεγκτές των προϋπολογισμών τους Ευρωπαίους και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο δίνεται επιχείρημα στους ευρωσκεπτικιστές τους Βρετανούς οι οποίοι λένε μα καλά γι' αυτό λέγαμε ότι δεν πρέπει να είμαστε μέσα στην Ευρώπη έχουμε καταφέρει να έχουμε μια λύση λούς-λούς ε, να μην είναι σαφής η κατάσταση κατά τρόπον ώστε να είμαστε όλοι σε ομοιρία Βέβαια ερώτηση δεν έκανα ακριβώς αλλά θα βρείτε τι θα απαντήσετε Ευχαριστώ κύριε Μοράλης Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε. Μέχρι τις 23 Ιουνίου φαντάζομαι ότι κάποια απάντηση θα σας δώσουν μέσω του τύπου της Βρετανίας. Ο κύριος Άζελμαν όταν έρθει η σειρά του θα μας απαντήσει ασφαλώς. Σίλβια Κάουφμαν. Αν θες να απαντήσεις. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και πολύ σύντομα. Θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και στο πλαίσιο του Eurojust σε λίγο. Έχουμε να κάνουμε μια περίπλοκη, ε, ένα περίπλοκο πλέγμα σχέσεων και βλέπουμε και στο Συμβούλιο ότι όταν συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε, είχαν γίνει διμερείς ε, συμφωνίες για να συναυθεί μια συμφωνία συνεργασίας με τη Eurojust. Και αυτό θα έχει το ρόλο του ασφαλώς. Στα όσα ανέφερε η κυρία Σπινέλη. Εγώ δεν λέω ότι πρόκειται για επιστοδρόμηση, αλλά για μία τάση να γίνουν πιο περίπλοκες οι προτάσεις σε σχέση με αυτό που αρχικά είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ότι αισθάνθηκε μεγάλη αμηχανία στην οικοδόμηση ενός τέτοιου ε, πλέγματος αρμοδιοτήτων. Εάν δηλαδή θέλουμε αυτό το νέο όργανο ο νέος θεσμός αυτός που θα θεσπιστεί να είναι σε θέση να αναλάβει δράση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτελεσματικότητα φυσικά. Εάν το θέλουμε αυτό πρέπει να έχουμε απολύτως σαφείς ορισμούς για την καθήλια αρμοδιότητα και όλα τα υπόλοιπα. Ιδάλλως, όντως, όπως είπε η κυρία Σπινέλη, κινδυνεύουμε να δούμε όπιστο δρόμο σε για πρόοδο. Και βέβαια δεν έχουμε περιθώριο ούτε καν πολιτικά να χάσουμε, να επιτρέψουμε να χαθούν χρήματα των τον Ευρωπαϊκό προπολογισμό, χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Πρέπει να αναλάβουμε από κοινού αποτελεσματικά βήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φράνσιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Ματέρα. Ξέρετε, οι Ολλανδοί είναι πρωταθλητές στη διαφάνεια. Η απάντηση είναι όχι δεν να συζητήσει στο Συμβούλιο επί του συγκεκριμένου θέματος. Πάντα τι υποτίθετο ότι ήταν αλληλένδετα τα δύο θέματα. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη στιγμή όπου οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ε, οριμάσει όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή και να δούμε αν θα υπάρξει ομοφωνία μεταξύ των 25 εκατών μελών αρχικά και θα δούμε μέχρι ποιου βαθμού θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις επί του ΠΙΦ αυτή είναι η απλή απάντηση στην ερώτησή σας. Η κυρία Αλεξάνδρα Τζιουρ Σρέντερ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να δώσω απάντηση. Κυρία Σπινέλη, εστιάζεστε βασικά στην ανάγκη να είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανεξάρτητο φορέα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κρίσιμο πυλώνα αυτό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν φορέα που θα λειτουργεί ανεξάρτητα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διάφορα μέτρα διαφύλαξης για να το εξασφαλίσουμε αυτό. Με, την, με το διορισμό πρώτα απ' όλα εκείνων που θα εργάζονται στο κεντρικό γραφείο και δεν θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών. Εδώ δεν είναι Eurojust, θα πρέπει ε, να είναι ανοιχτό στους εισαγγελείς και θα πρέπει να εγγυηθούμε ανεξαρτησία σε αυτούς και θα υπάρχουν και άλλα μέτρα διαφύλαξης στο κείμενο, όπως η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους διάφορους φορείς στην, κεντρικό, στην κεντρική υπηρεσία και θα δώσουμε ευρωπαϊκή υποστηθέμενη αξία του το τρόπος. Δίκιο έχετε, είναι βασικό θέμα για μας. Πρέπει να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία της ΕΠΟ. Να είναι εξάρτητη η διοκτική αρχή. Όσον αφορά την κυρία Ζίπελ, αν πρέπει να ζητάει εισαγγελία, ευρωπαϊκή εισαγγελία από τα κράτη-μέλη, τον αναλάβει τις υποθέσεις δεν φτάσαμε εκεί. Θα υπάρχουν μηχανισμοί και ο κανονισμός εμπεριέχει διάφορες υποθέσεις και περιπτώσεις και προβλέπει και υποχρεώσει των κρατών μελών να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή ότι υπάρχει κάποια υπόθεση. Όπως είπα και στη δήλωσή μου, αποκλειστική αρμοδιότητα θα απέφευγε αυτά τα προβλήματα. Αλλά αν ο κανονισμός προβλέπει επαρκείς κανόνες περί καθηκόντων και σωστά είπε ο Νίκολας ότι ήδη θα έχει κατά προτεραιότητα κάποιες αρμοδιότητες. Αυτό είναι ένα καλό βήμα για το δεύτερο που είπατε. Πώς αποφεύγουμε ε, κάποιο να επιδιώκει κάποιος να βρει την πιο εύκολη, τον πιο εύκολο φορέα για να προωθηθεί μια υπόθεση. Θα πρέπει να βρούμε μηχανισμό το, σύμφωνα με τον οποίο θα καθορίζεται το αρμόδιο δικαστήριο ε, η κυρία Γκρέσλε ρώτησε τι κάνουμε για την νομική βάση. Καταρχάς σας έχουμε την έγκριση της οδηγίας PIF. Θα χαιρόμουν να το έβλεπα αυτό. Και μετά αναλύουμε λεπτομερώς κατά πόσο θα πρέπει να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή όχι. Δεν έχω απάντηση σήμερα. Όμως θέλω να πω στο ακροατήριο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το άθρο 325 ως νομική βάση. Δεν το κάναμε αυτό διότι ε, το ήθαν τα κράτη-μέλη, διότι προβλέπεται αυτή η νομική βάση στη συνθήκη που αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το άθρο 325 και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπεριλαμβάνεται και το ποινικό δίκαιο. Και ήταν λογική προσέγγιση μας. Το τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες ε, θα το δούμε. Το αφήνουμε ανοιχτό για την ώρα. Καλώς, τελειώσαμε. Ευχαριστώ για μία σύντομη παρουσίαση, άκρος ε, περιεκτική. Στο δεύτερο τμήμα της Ακράσος πάμε στον Άξελ Βος που θα προεδρεύσει αυτού του τμήματος που συντάσσει ε, το σχέδιο κανονισμού για το Eurojust. Παρακαλώ να έρθει εδώ μαζί με τους ομιλητές. Μισελ Κόνιξ, πρόεδρο της Eurojust, Τζοβάνι Κέστερ, γενικό διευθυντή της Όλαφ. Παρακαλώ να έρθετε εδώ, στο Εδράνο. So, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Καλώς ορίσατε λοιπόν όλοι για το δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Η κυρία Μισελ Κόνιγκς είναι εδώ πρόεδρος της Eurojust, κύριος Κέσλερ. Αυτό είναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Από την Ούλαφ. Και Ξεκινώ αμέσω. Με τα θέματά μας βεβαίως είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορεί πέραν της Eurojust να αναπτυχθεί και η ΕΠΟ. Έχουμε μερικές φορές την εντύπωση ότι θα υπάρξουν δύο ανεξάρτητα όργανα εδώ όπως τουλάχιστον έχει σχεδιαστεί μέχρι τώρα το σύστημα. Σε σχέση με το άρθρο 3, παραγραφος 3 του κανονισμού ΕΠΟ και το άρθρο 57.6 της συνθήκης αποκόπτεται και αναπτύσσεται χωριστά από τη Eurojust. Το ΕΠΟ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή ανεξάρτητα αλλά στενά συνεργαζόμενα όργανα λοιπόν. Και θα αναλάβει νέα καθήκοντα τι εισαγγελία, δηλαδή η ΕΠΟ. Και βέβαια καθήκον μας είναι όλα τα κρατημέλη να το υποστηρίξουμε. Κυρία Κόνιγκς τώρα. Παρακαλώ να λάβει το λόγο για να μας κάνει την παρουσίασή της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου δίνετε τη δυνατότητα να τονίσω τη σημασία του μελλοντικού κανονισμού για τη Eurojust και την εξίσου μεγάλη σημασία άλλων κανονισμών και συγκεκριμένα του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για μια σημαντική χρονική στιγμή. Το μέλλον της Eurojust ε, είναι άκρο σημαντικό για μας όπως καταλαβαίνετε και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, αρχικές παρατηρήσεις. Έχουμε δουλέψει με τα κράτη-μέλη, για τα κράτη-μέλη ε, και έχουμε νομίζω καταφέρει να ναι. προχωρήσουμε με το επιχειρησιακό έργο αλλά και με τις συγκεκριμένε πολιτικές, δηλαδή το οικοδόμηση δικτύων για διάφορα ζητήματα που ενδιαφέρουν στο ευρύτερο πλαίσιο της ασφαλείας ε, δικαίου. Και η έμεση απόδειξη του ότι προχωρούμε είναι ότι έχουμε περισσότερες ε, ε, συνεδρίες συντονισμού, περισσότερες ευνητικές ομάδες, περισσότερες υποθέσεις, άρα όλα αυτά αποδεικνύουν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην Eurojust. Η Eurojust παρά τα διαφορετικά νομικά συστήματα, χωρίς ιδιαίτερη εναρμόνιση, κατάφερε να ε, εξασφαλίσει ε, την επιτάχυνση ε, της δικαστικής ενεργασίας και να βελτιώσει το συντονισμό. Θέλω να ευχαριστήσω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο ιδιαίτερος για την πολύ καλή τους δουλειά στον κανονισμό περί Ευρωπόλη. Αυτό έχει σημασία γιατί σίγουρα και το πώς αντιδρά η αστυνομία επηρεάζει και τον κανονισμό της Eurojust. Αν θεωρεί κανείς ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο, τη διακίνηση ανθρώπων μόνο από την ε, αστυνομία αφήνοντας ε, τελείως εκτός ε, τη δικαστική συνέχεια που δίνεται, δεν πρόκειται να έχει την επιτυχία. Το τονίζω και αυτό λοιπόν και βέβαια τονίζω και τη σημασία Μία πολύ σαφού διασύνδεσης μεταξύ Eurojust και Γραφείου Ευρωπαϊκού Αγγελέα. Άρα, για να περάσω σε αυτές τις αρχικές παρατηρήσεις, όπως είπα, κάναμε πολλά και ό,τι γίνει με οποιοδήποτε κανονισμό, όλα αυτά πρέπει να μας δίνουν τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τις ε, δυνατότητες μας ακόμη περισσότερο. Ό,τι και αν γίνει σε άλλους κανονισμούς θα πρέπει να γίνει με συνεκτικότητα, με συμμετρικό και συμβατό τρόπο και όχι αντιφατικό. Αυτό είναι το πρώτο, το προκαταρκτικό μου σχόλιο. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι τελικά αναγνωρίζουμε το έργο, ε, το σκληρό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Και καταρχήν επικροτούμε τη γενική προσέγγιση του Μαρτίου 2015 του Συμβουλίου. Γιατί ε, είναι νου στο Συμβούλιο στις προτάσεις και τις ανησυχίες της Eurojust. Εξού και επικροτούμε την αρχή και τις αλλαγές τις οποίες προτείνει το Συμβούλιο. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά σημεία που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας για να μην χάσουμε την ευκαιρία να είμαστε αποτελεσματικοί υπό την οπτική γωνία τουλάχιστον της Eurojust. Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Eurojust, την πρόταση της Κομισιόν για την ουσιαστική αρμοδιότητα είναι μειωμένες οι αρμοδιότητες μας σε σχέση με τώρα. Υπάρχει ένα παράρτημα στον κανονισμό με τον κατάλογο των αξιόπινων πράξεων. Στο άρθρο 3 προτείνεται η προσθήκη μιας νέας παραγράφου για την αρμοδιότητα της Eurojust για τύπους αδικημάτων πέραν αυτών που καταγράφονται. Κατόπιν δήματος της αρμόδιας αρχής. Θα θέλαμε να ισχύσει αυτό και στο μέλλον. Θέλουμε ευελιξία. Υπάρχουν νέες μορφές αξιόπινων πράξεων και αδικημάτων. Όλο και πιο πολύπλοκα γίνονται τα αδικήματα, άρα και εμείς θα πρέπει να είμαστε στην αιχμή Θέλουμε λοιπόν η ευέλικτη προσέγγιση που να διατηρεί και το status quo. Τώρα, πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει δεν υπάρχει αρμοδιότητα της Eurojust για τα δικήματα τύπου PIF, όπως λέγονται, στα οποία είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διάταξη αυτή δεν είναι ευθυνωσμένη με άλλες ε, διατάξεις και στο παράρτημα 1 που υπάρχει ένας κατάλογος αναφέρεται το ΠΙΦ. Άρα πρέπει να διευκρινιστεί το άρθρο 3, ότι δεν συνάδει με τις άλλες διατάξεις. Πρέπει να διασταυρώσετε τι λέει και στην ε, βερσιό του κειμένου της ε, ε Κομισιόν που μιλά για exclusive competence. Πρέπει να διευκρινιστούν αυτά. Εμείς εστιάζουμε στη σημασία, στο χαρτοφυλάκιό μας, να έχουμε αρμοδιότητα και για αυτά τα θέματα. Άρα πρέπει να διευκρινιστεί. Άρθρο 3 σε σχέση με το παράρτημα και τον κατάλογο. Τώρα, γενικά θεωρούμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια, μεγαλύτερη ευελιξία, τα κράτη-μέλη έχουν πλέον την εξουσία στα χέρια τους. Έχουμε και μια πολύ καλοδεχούμενη παράγραφο, την παράγραφο 8, που λέει για εκχώρηση περαιτέρω ε, αρμοδιοτήτων που δεν προβλέπονται στον κανονισμό. Άρα μεγαλύτερη ευελιξία προς ανατολισμένους επαγγελματίες του κλάδου. Επίσης, ό,τι αφορά την κυβέρνηση της Eurojust, θεωρούμε ότι το κείμενο αντιμετωπίζει και διασκεδάζει τις ανησυχίες μας και είναι καλό. Κάτι άλλο σημαντικό που έχει να κάνει με τη Eurojust και τη Europol και συγκεκριμένα δύο σημεία θέλω τώρα να αναφέρω. Το πρώτο αφορά την ιδέα της Κομισιόν για εφαρμογή της αρχής αμοιβαιότητας στην ανταλλαγή πληροφοριών. Χαιρόμαστε που στόχος είναι η ομαλή ε, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Γιώργης και Europol παραμένουν και στους δύο κανονισμούς. Βέβαια, ακόμη και στη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, το κείμενο δεν εφαρμόζει την αρχή της αμοιβαιότητας. Και αυτό δεν εφαρμόζεται ως αρχή ισότιμα στη Europol και στη Eurojust. Άρα και στους δύο κανονισμούς, Eurojust και Europol, πρέπει να υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης ε, του ε, οργανισμού, αλλά αυτό επιβάλλεται προς το παρόν μόνο στη Eurojust και όχι ε, στη Europol. Θα έπρεπε λοιπόν να τροποποιηθεί το άρθρο 40 του σχεδίου κανονισμού. Ανταλλαγή πληροφοριών λοιπόν βάσει της αμοιβαιότητας και από τις δύο πλευρές όμως. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του G, τώρα ξέρετε ότι 11 Μαρτίου ε, αποφασίστηκε θα είμαστε υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση και εμείς. Ε, καλό είναι αυτό. Δύο οργανισμοί να είναι αρμόδια για τη χρηματοδότηση JIT. Ίσως όμως υπάρξουν κάποιες αλληλεπικαλύψει, ε, διπλή χρηματοδότηση, κάποιες παρανοήσεις. Λέγεται ήδη στο κανονισμό Europol θα πρέπει να θεσπιστούν όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή και οι σχετικές διατάξεις κανονισμού Europol και του σχεδίου κανονισμού Eurojust πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση και πρέπει ε, η μία, ο ένας κανονισμός να αντικατοπτρίσει στον άλλο. Ελπίζουμε αυτό να ε, συμβεί και στο τελικό κείμενο. Πέραν τη ευθυγράμμιση των σχετικών διατάξεων, θα χρειαστεί και ένα μηχανισμό συντονισμού. Καλό είναι να έχουμε όρου, προποθέσει, ένα μηχανισμό κτλ. Όμω, απαιτείται ο μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των δύο οργανισμών, ώστε και στην πράξη να εξασφαλίζεται αυτή η συνεκτικότητα και η συνέπεια. Και για τη γραμματεία του δικτύου JIT, που έχει πολλή εμπειρία συχνά και τακτικά συνεργάζεται με την Europol και αυτή η γραμματεία θα μπορούσε πραγματικά να διευκολύνει τον συντονισμό, να μην επανεφεύρουμε τον τροχό. Έχουμε τις εμπειρίες μας, μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτές. Και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τη σημαντική διασύνδεση Eurojust και Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Η σχέση των δύο αυτών φορέων θα ήθελα να τονίσω είναι σημαντική, αλλά οι δύο φορείς είναι ξεχωριστοί, είναι ανεξάρτητοι. Είπαμε και τονίζουμε ότι οι γερόντζες θα πρέπει να αρμοδιότητες για τα δικήματα πιφ, το ξανά από αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα το κείμενο του κανονισμού περί εισαγγελίας θα είναι δύο διαφορετικές οντότητες, Eurojust και Ευρωπαϊκή Σικελία, που θα συνεργάζονται μεταξύ τους όμως, θα έχουν διασύνδεση με επιχειρησιακούς, διαχειριστικού δεσμούς. Παρά την ερμηνεία του άρθρου 86, πρέπει να οριστούν σαφείς δεσμοί, να είναι ξεκάθαρη η διασύνδεση των δύο φορέων. Ναι, μεν υπάρχει, είναι σαφές αυτό, ότι θα υπάρχει σχέση μεταξύ Eurojust και ΕΠΟ, ε, Ευρωπαϊκή αλλά θα πρέπει σε επίπεδο ε, επιχειρησιακό και διαχειριστικό να ε, διευκρινιστούν επαρκώς αυτές οι διασυνδέσεις. Τώρα η σχέση των δύο αυτών φορέων περιλαμβάνει υποχρεώσει και δικαιώματα για τις δύο πλευρές. Eurojust και Ευρωπαϊκή Αγγελία, για παράδειγμα, θα πρέπει να έχουν αμοιβαία καθήκοντα. Δηλαδή να ενημερώνουν οι μεν τους δε. Μιλάμε ουσιαστικά για αμοιβαίο σεβασμό και δικαιοσύνη. Και σίγουρα θα πρέπει να αποφεύγεται η ε, διπλή ερμηνεία. Συμμετρική, συμβατική κανόνες. Μία αντιφατική και όπως είπα να αντικατοπτρίσει το ένας κανονισμός στον τρόπο στον άλλο. Τέλο, η Eurojust ε, είναι διατεθειμένη να στηρίξει τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Αγγελία. Όλοι άλλωστε οι οργανισμοί πρέπει να συνεργάζονται σε καιρού λιτότητα και ανευπροηγουμένων προβλημάτων στον τομέα τη ασφάλεια και απειλών για την ασφάλεια. Θα πρέπει να ενώσουμε τι δυνάμει μα να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε και πράγματι θα βάλει και η Eurojust το λιθαράκι της για να βοηθήσει στη δημιουργία Τη Ευρωπαϊκή Έγκυρης. Συγκεκριμένα όμως, εάν η Eurojust να λάβει νέα καθήκοντα, θα χρειαστεί και ενό πόρου, έτσι. Είναι σαφέ αυτό. Και θέλω να τονίσω ότι η Eurojust δεν θα στηρίξει διακανονισμού όπου ενδεχομένω ε, περιοριστούν μέσω αυτών οι Δικαιοδοσίε μας ε, και οι αρμοδιότητέ μας. Ναι, με να συμβάλλουμε, αλλά ποτέ σε βάρος των υπηρεσιών που στηρίζουν τη βοήθεια που παρέχουν. Και επαναλαμβάνω κυρίω εν καιρό κρίση. Όπω όπως βλέπετε στη διαφάνεια έχουμε με άνευ προηγουμένου κρίση στον τομέα τη ασφάλειας και πέρσι πάνω από 23%. Πάνω από 23% ήταν η αύξηση των υποθέσεων οι περισσότεροι αφορούσαν την καταπολέμηση τρομοκρατίας, ε, το κυβερνοέγκλημα, τη, τη διακίνηση ανθρώπων, λαθρεπό κτλ. Εμείς είμαστε τεθειμένοι να συνεργαστούμε και πρόθυμοι να συνεργαστούμε, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε όλο και περισσότερες δυνατότητες και αρμοδιότητες και όχι λιγότερες. Και αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί και στον κανονισμό ΕΠΟ και στον κανονισμό Eurojust. και αν έχουμε, επαναλαμβάνω, νέα καθήκοντα, θα πρέπει να έχουμε και νέε δημοσιονομικέ ρυθμίσει για να έχουμε του απαιτούμενου πόρου, τα απαιτούμενα μέσα στη διάθεσή μα. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ για την ε, εστιασμένη αυτή προσοχή στα θέματα Βεβαίως, πέραν της Europol υπάρχει και η Όλαφ. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε, οι δυνατότητες που υπάρχουν. και οι σχέσεις μεταξύ των αρχών αυτών. Παρακαλώ κύριε Κέσλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και την Επιτροπή σας για την πρόσκληση και την ευκαιρία να σας μιλήσω στο Ευρωκοινοβούλιο για το σημαντικό αυτό θέμα με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αλλάζει το τοπίο κατά πολεμήσεως των απατών και επιθέσεων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν είναι απλή μεταρρύθμιση. Το τοπίο θα αλλάξει. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ΕΠΟ που θα είναι ερευνητικός και διεκτικός φορέας να βασίζεται σε άλλους υφισταμένους φορείς την Όλαφ που είναι ο μόνος οργανισμός ερευνητικό Ευρωπαϊκή Ενώσεως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και ναι βασίζεται και στο Eurojust, που όπως υπόθηκε είναι ο μόνος ευρωπαϊκός δικαστικός οργανισμός. Άρα, θα ήταν εσφαλμένο εξ αρχής αν δεν θεωρήσουμε αυτή τη βασική αλλαγή του θεσμικού περιβάλλοντος ως κάτι περίπλοκο και πολυσχηδές που πρέπει να ληφθεί συνολικά σφαιρικά υπόψη. Το Συμβούλιο το συζήτησε το θέμα αυτό σε επίπεδο ομάδα εργασίας. Και κάποιες διατάξεις για τα ζητήματα αυτά ήδη έχουν συνταχθεί. Θα υποβληθούν στο Συμβούλιο του Ιουνίου για έγκριση. Εμείς σαν Όλαφ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουμε τα μέτρα τα κράτη-μέλη πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις σχέσεις μεταξύ των τριών φορέων. Και πιστεύω ότι οι διατάξεις που διέπουν τις σχέσεις ΕΠΟ και Όλαφ πετυχαίνουν σωστή ισορροπία. Με κάποιους όρους στα πλαίσια του μοντέλου για την ΕΠΟ που έχουν επιλέξει τα κράτη-μέλη. Γιατί το λέω αυτό. Και ερχόμαστε εδώ στην πρώτη διαφάνεια για να καταλάβουμε και να πάρουμε απόφαση για τη σχέση μεταξύ των τριών φορέων πρέπει να ξεκινήσουμε από την ερώτηση που συζήτησε το προηγούμενο πάνελ που είναι θεμελιώδη σημασία. Τι είδους έπο θα έχουμε, τι αρμοδιότητες θα έχει ο φορέας αυτός και από εκεί θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση με τους υφιστάμενους φορείς και οργανισμούς. Λοιπόν, με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο υπενθυμίστηκε, η Ευρωπαϊκή Αγγελία θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για αδικήματα πιφ. Σημαντικότατο ζήτημα αυτό. Ξέρουμε ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Συζητήθηκε από το προηγούμενο πάνελ το θέμα αυτό. Ήταν αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποιες εξαιρεσει από τι αρμοδιότητε της Ευρωπαϊκής Εισαγγελική Αρχής στα δικήματα ΠΙΦ και η ΕΠΟ θα μπορεί να ερευνά μια υπόθεση αν η ζημία που έχει προκληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά τη ζημία που έχει προκαλέσει, προκληθεί σε άλλο θύμα. Το Συμβούλιο έχει εισαγεί κάποια κριτήρια που πιστεύω ότι είναι ανησυχητικά. Συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε. Κριτήρια λέγω τα οποία από τη μία πλευρά θα αποκλείουν τεράστιο αριθμό υποθέσεων πιφ από τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από την άλλη πλευρά με την εισαγωγή κάποιων κριτηρίων τα οποία κατά την άποψή μας βάσει της εμπειρίας της Όλαφ θα είναι κριτήρια δύσκολα να ερμηνευθούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις και θα είναι κριτήρια δύσκολο να εφαρμοστούν και θα υπάρχει ο κίνδυνος συγκρούσος μεταξύ Ευρωπαϊκής Αγγελίας και εθνικών δικαστικών αρχών. Άρα, σε όλες τις υποθέσεις και περιπτώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που συζητούνται στο Συμβούλιο, η αρμοδιότητα θα είναι κοινή και θα μοιράζεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κρατών μελών. Αρκετά περίπλοκη είναι η κατάσταση. Απ' τη μία πλευρά θα αφήσει πολλές, πολλές υποθέσεις πιφ εκτός αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και σε άλλες περιπτώσεις θα υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων και θα δημιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πού βρισκόμαστε εμείς ως Όλαφ. Καταρχάς έχουμε περιθώριο να υπάρχουμε, χώρο. Πρέπει να δούμε και πώς θα αντιμετωπιστούν τα κράτη-μέλη που δεν θα συμμετέχουν στην ΕΠΟ και με τις υποθέσεις εκτός αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αγγέλιας. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Πρέπει να ξεκινήσουμε από δύο βασικές αρχές που αναφέρονται στον κανονισμό για τη σχέση μεταξύ Όλαφ και ΕΠΟ στην περίπτωση της Όλαφ, λόγω του ρόλου που διαδραματίζει σε διοικητικές έρευνες, είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεται με την ΕΠΟ και θα πρέπει να κρατήσει η Όλαφ την αρμοδιότητά της στα δικήματα ΠΙΦ για υποθέσεις που θα εξετάζονται αποκλειστικά από τα κράτη-μέλη. Οι δύο βασικές αρχές λοιπόν είναι ότι παράλληλες έρευνες Όλαφ και ΕΠΟ θα πρέπει να αποφεύγονται. Δεν θέλουμε ε, διπλή δουλειά, επικάλυψη, αλληλεπικάλυψη. Όταν ξεκινά η ΕΠΟ την έρευνά της, η Όλαφ δεν θα έχει αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη έρευνα, δεν θα ερευνά το ίδιο θέμα, εκτός αν ζητηθεί κάτι τέτοιο από πλευράς ΕΠΟ που χρειάζεται υποστήριξη. Δεύτερον, ακόμα και αν η ΕΠΟ έχει ξεκινήσει μια έρευνα ή σε περιπτώσεις όπου θα μπορούσε να ξεκινήσει έρευνα η ΕΠΟ υπάρχει περιθώριο για διοικητική έρευνα που διενεργεί η Όλαφ. Διοικητική έρευνα καμιά φορά είναι χρήσιμη σαν προπαρασκευαστικό βήμα για έρευνα στον εγκληματικό τομέα, στον ποινικό τομέα. Μπορεί να παίξει ένα συμπληρωματικό ρόλο. Συνέχεια και ανάκτηση, οικονομική ανάκτηση ποσών. Ε, μπορεί να παίξει ρόλο η Όλαφ, η ποινική διαδικασία δεν μπορεί να το καλύψει αυτό το θέμα με τον ίδιο τρόπο. Ας πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Έχουμε δύο περιπτώσεις όταν η ΕΠΟ δρά ε, για μια συγκεκριμένη υπόθεση και τη δεύτερη περίπτωση που δεν δρά, δεν κινείται. Όταν λοιπόν η ΕΠΟ αναλάβει μια υπόθεση και την επεξεργάζεται, σε αυτή την περίπτωση η Όλαφ πάντα μπορεί να δράσει σαν πηγή πληροφοριών για ενδεχόμενα δικήματα ΠΙΦ που θα πρέπει να διαβιβαστούν στην ΕΠΟ ούτω ώστε να διεξαγάγει τις δικές της έρευνες. Έχουμε ένα ευρύ δίκτυο, παγκόσμιο δίκτυο, συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με ιδιωτικούς πόρους, πηγές που μας επιτρέπει να συλλέξουμε 1.400 πληροφορίες το χρόνο για δικήματα PIF που όταν χρειάζεται θα μπορούσαν να προωθηθούν προς την ΕΠΟ για να ξεκινήσει έρευνα για ποινικά δικήματα, όπως κάνουμε τις εθνικές αρχές σήμερα. Δεύτερον, όταν η ΕΠΟ επεξεργάζεται μια υπόθεση, μπορεί η Όλαφ να υποστηρίξει τις έρευνες ΕΠΟ μέσω αναλύσεως, τεχνογνωσίας, επιστημονικών μεθόδων και να διαθέτουμε και το δίκτυο που διαθέτουμε με τις, ε, που συμμετέχουν οι εθνικές υπηρεσίες. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν η ΕΠΟ δεν αναλάβει μια υπόθεση, λόγω περιορισμένων αρμοδιοτήτων αυτής, η Όλαφ υπέχει καθήκον να διενεργήσει τις δικές της έρευνες, όπως κάνουμε σήμερα. Θα ήταν παράδοξο αν με τη θέσπιση της ΕΠΟ έχουμε λιγότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων στα κράτη-μέλη που, παραδείγματος χάρη, δεν θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή σε τομείς όπου η σε τομεις που Εισαγγελία δεν καλύπτει λόγω περιορισμένων αρμοδιοτήτων. Η ΕΠΟ μπορεί να ενημερώνει την Όλαφ για περιστάσεις κατά τις οποίες η ΕΠΟ δεν ξεκινά έρευνες ή αν α, απορρίψει μια υπόθεση. Εν κατακλείδη λοιπόν πιστεύω ότι η ΕΠΟ και η ΟΛΑΦ έχουν μια σχέση που βασίζεται στην πληρωματικότητα των εντολών των δύο φορέων και μπορεί να απορρέψουν μόνο καλά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της απάτης και επιτρέψτε μου να πω και να αποφύγουμε λόγω συμπληρωματικότητας των δύο σωμάτων αυτών να αποφύγουμε λέγω κάποιες ζημίες που προέρχονται από τον περιορισμό της εντολής που θα έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λόγω αυτών των περιορισμών ανοίγουν κάποια κένα που μπορούν να καλυφθούν λόγω της συμπληρωματικότητα των δύο αυτών φορέων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε και για την παρέμβασή σας. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να διατυπώσουμε ερωτήσεις. Εάν δεν είστε κανείς το λόγο, θα ήθελα εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Βεβαίως, Τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καταπολέμηση των, του εγκλήματος στον τομέα αυτών είναι ο στόχος μας. Ακούγοντας τις τοποθετήσεις σας, βλέπω ότι υπάρχει έλλειμμα ως προς τις αρμοδιότητες Eurojust, Olaf, ΕΠΟ και εθνικές αρχές συνιστούν ένα πολύ περίπλοκο πλέγμα. Και ναι, φαντάζομαι ότι θα κάνετε κάποια διαφοροποίηση, ίσως ο καθένας από την σκοπιά του, αλλά θέλω τις απόψεις. Γιατί νομίζω ότι όταν έχουμε να κάνουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, δεν ε, βοηθάει να τα αφήνουμε σε ένα τόσο περίπλοκο μπλέγμα. Νομίζετε ότι η ΕΠΟ και η Eurojust, παραδείγματι, θα μπορούσαν να υπολογίσουν κάποια περίπτωση στην οποία θα μπορούσε να γίνει μια ε, διάκριση αρμοδιοτήτων που θα επέτρεπε ταυτόχρονα και τη συνεργασία. Και δεύτερον, εμείς ως νομοθέτες θα μπορούσαμε ενδεχομένω να σκεφτούμε την ε, υπαγωγή αρμοδιοτήτων για την καταπολέμηση της, ε, του οικονομικού εγκλήματος της Όλαφ ε, σε ένα βαθμό τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό θα σήμαινε όμως αποστέρηση κάποιων τέτοιων εξουσιών από την ίδια την Όλαφ. Οπότε τι θα έμενε ως αρμοδιότητα της Όλαφ. Αν προχωρούσαμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι το ερώτημα και το πιο δύσκολο βέβαια είναι το θέμα της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές. Εκεί όπου η ΕΠΟ δεν αναλαμβάνει δραστηριότητα έχω την αίσθηση ότι είναι πολλές οι υπηρεσίες οι οποίες αναμονίονται στην καταπολέμηση των αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να τα να διαρθρώσουμε, να ξεχωρίσουμε, να οργανώσουμε αυτές τις ε, αρχές και τις αρμοδιότητες τους. Έχετε κάτι να προτείνετε εδώ και ρωτώ αν υπάρχει και άλλη ερώτηση από τους συναδέλφους. Λοιπόν, Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ναι, μιλούμε για ποινική δικαιοσύνη ουσιαστικά. Πρόκειται για ένα θεμελιώδου σημασία ζήτημα. Υπάρχουν δύο θεωρήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ουσιαστικά χαρακτηρίζουν τη συζήτησή μας. Ένας πρώτος τρόπος ε, να χαρακτηριστεί η ποινική δικαιοσύνη θα ήταν να πει κανεί ότι ανήκει αποκλειστικά στα κράτη-μέλη και άρα θα υπάρξει μόνο μια χαλαρή συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών, όχι σε μια Ευρώπη των εθνών, η οποία έτσι θα προσλαμβάνει το νόημά τη, αλλά είναι προφανέ ότι δεν πρόκειται για το μοντέλο και ότι εγώ το θεωρώ ω το πιο αποτελεσματικό το οποίο έχει επιλεγεί. Και το δεύτερο είναι αυτό της ολοκλήρωσης, της ενοποίησης, δηλαδή πέραν των εθνικών δικαστικών αρχών, ποινικών δικαστικών αρχών, θα εγκαθιδρυθεί μια ευρωπαϊκή ποινική δικαιοσύνη. Είναι σαφές από τη συζήτηση για το σημερινό θέμα, αυτό το θέμα της ΕΠΟ δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα από ό,τι στο παρελθόν και βέβαια εδώ και ότι είναι σαφής ο πολιτικός στόχος, πιο ενοποιημένη και πιο ομοσπονδή Ευρώπη. Ε, αυτό, αυτή είναι η λογική που οδηγεί προς τις επιλογές αυτές, αλλά καθιστά ταυτόχρονα και πολύ πιο περίπλοκο αυτό το σύστημα και από τα όσα ακούω σήμερα, πολύ φοβούμαι ότι θα είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα και άρα δεν θα μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Ε, δύο τύποι συγκρούσεων νομίζω ότι είναι πιθανό να αναδειχθούν. Σύγκρουση αρμοδιότητα μεταξύ ΕΠΟ και κρατών μελών, γιατί θα είμαστε σε συντρέχουσα αρμοδιότητα, σε συντρέχουσες αρμοδιότητες και όπως είπε και ο κύριο Κέσλερ, είναι προφανώς ότι θα προκύψουν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και δεύτερον, δεύτερο πρόβλημα το οποίο θα εμφανεί ίσως και πιο ε, γρήγορα, πιο νωρίς, γιατί το βλέπουμε ήδη να διαφαίνεται, σύγκρουση μεταξύ ΕΠΟ και Όλαφ. Η Όλαφ ως υπηρεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης έχει συγγενική με τις ΕΠΟ ε, συγγενικές με τις ΕΠΟ αρμοδιότητες, γιατί στόχος της είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Η περίφημη ΠΙΦ δεν αφορά μόνο την ΕΠΟ, αφορά και την ε, Όλαφ. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ, μήπως τελικά η ύπαρξη της ίδιας της Όλαφ θα τίθεται ένα αμφιβόλο με την ε, σύσταση αυτής της ΕΠΟ για τους δύο αυτούς λόγους που ανέφερα, δηλαδή τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων, πρώτα απ' όλα γιατί ο ένας από δύο θα περισσεύει και δεύτερον γιατί η Όλαφ είναι οργανισμός που έχει χάσει την αξιοπιστία του. Έχω διαβάσει εκθέσεις που κάθε άλλο παρά εγκομιαστικές είναι. Αυτή ήταν η ερώτησή μου, κυρία Κέσλερ. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις άλλες. Όχι από ό,τι βλέπω. Και για παρα... γι' αυτό παρακαλώ να προχωρήσουμε σε απαντήσεις. Η κυρία Κόνη και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις Σα Μπορώ να συνδυάσω τις δύο ερωτήσεις θα απαντήσω αγγλικά. Αρχική ιδέα το άρθρο 84 και το άρθρο 86 της Συνθήκης Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ήταν κάτι σαφές. Η Eurojust ήταν οριζόντιος οργανισμός και όλες οι προσπάθειες έπρεπε να καταβληθούν ούτως ώστε να ο οριζόντιος φορέας να είναι ενισχυμένος. Θέλαμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες της Eurojust. Για κάποιο λόγο αυτό το άρθρο το 85 στην προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρήθηκε ότι είναι μια εξέλιξη αλλά όχι επανάσταση. Οριζόντιο είναι καλό, όπως εξήγησα, μπορεί να υπάρχει διασύνδεση με τα κράτη-μέλη, χωρίς μεγάλο βαθμό εναρμόνισης οικοδόμηση εμπιστοσύνης ε, μέσω συντονισμού και συνεργασίας. Ο συντονισμός και η συνεργασία θα μπορούσαν να ενισχυθεί με κάποια σημεία μέσω του άρθρου 85-86 αφορούσε μία κάθετη ολοκλήρωση και θέλαμε να εστιαζόμεθα επί συγκεκριμένου τομέα ε, αδικημάτων και κλιμάτων, τομέα πιφ. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι μετά τις συζητήσεις και μετά την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά τις προσπάθειες του Συμβουλίου, ακόμα δεν ξέρουμε τι αντιπροσωπεύει ένα έγκλημα, ένα δίκημα πιφ. Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Προσεγγίσαμε όλα τα κράτη-μέλη, την Europol, την Olaf και έχουμε την πρακτική συμφωνία μεταξύ Olaf και Eurojust. Πρακτικό αποτέλεσμα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά το 2015 έχουμε καλά παράδειγματα. Έχουμε την ε, κοινή ερευνητική ομάδα με τη συνεργασία της Όλαφ για θέματα φοροαποφυγή, λαθρεμπόριο τσιγάρων, ξέπλυμα χρήματων, το σύστημα καταπολεμής του λαθρεμπορίου τσιγαρέτων, Είχαμε παραγωγή σιγαρέτων που εξήγονται μαζικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με παράδοξη παραγωγή. Συνεργαστήκαμε. Υπήρξε καλή συνεργασία 20 υποθέσεις, είχαμε 5 συντονισμούς σε επίπεδο Eurojust με πλήρη συμμετοχή της Όλαφ για το λαθρεμπόριο τσιγάρων που είναι αδίκημα πιφ. Όσον αφορά απάτη ΦΠΑ έχουμε ιστορικό υποθέσεων και συντονισμού και ομάδων, κοινών ομάδων ερευνητικών με συμμετοχή κρατών μελών, πολλών. Εάν κάνουμε κάποια προσπάθεια. Αν περάσουμε μέσω κανονισμού, η μόνιμη ανησυχία και ανησυχία του Τζοστ και όλων των κρατών μελών, των δικαστικών φορέων, των δικαστικών φορέων των κρατών μελών είναι η απλούστευση. Να είναι κάτι απλό και εύληπτο για τους ε, εισαγγελείς και τις οπτικές αρχές. Το κείμενο ως υπευλήθη, όπως είπε ο κ. Γκέσσερ, δημιουργεί κάποια ενδεχόμενα συγκρούσεων το γύρο Eurojust μπορεί να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή, έχει συνηθίσει. Αν έχει αρμοδιότητα όμως για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ παρακαλώ τον κύριο Κέσλερ να λάβει πάλι το λόγο. Εγώ δεν θέλω να κρατήσω ζωντανή την Όλαφ με κάθε τρόπο. πρέπει να ομολογήσω κάτι. Κυρίως απευθυνόμενος προς τους αμφιβάλλοντες. Μέχρι πριν ένα-δύο χρόνια θεωρούσα ότι όλα θα είχε πεθάνει και θα είχε σωματωθεί στην ΕΠΟ. Αυτή θα ήταν η σωστή λύση σε κάποιο βαθμό, με κάποια όρια. Δεν θα τα αναφέρω τώρα. Κατά κάποιο τρόπο ήταν αποτέλεσμα της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΠΟ. Κάτι στο οποίο συμβάλαμε και εμείς. Όπως είπα όμως, αν θέλουμε να μιλήσουμε περί συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων, πρέπει να ξεκινήσουμε από τις αρμοδιότητες αυτών. Δηλαδή, για τις αρμοδιότητες της ΕΠΟ. Τώρα έχουμε μία ΕΠΟ με πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες όσον αφορά τις υποθέσεις πιφ και με κανόνες οι οποίοι φοβάμαι και θεωρώ και ελπίζω να ασφάλω δύσκολο να ερμηνευθούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις και δύσκολο να εφαρμοστούν. Αυτό θα οδηγεί σε συγκρούσεις με τις αρχές των κρατών μελών. Βεβαίως, βεβαίως, όχι με την Όλαφ. Και η Όλαφ εφόσον μιλάμε για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, εφόσον είμαστε στο ίδιο καράβι και όλοι νοιαζόμαστε γι' αυτό, σε αυτή την περίπτωση με τόσο περιορισμένες αρμοδιότητες που δίδονται στην ΕΠΟ για την έναρξη ποινικών ερευνών για εγκλήματα πιφ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο υπάρχει μεγάλη ανάγκη θα έλεγα διοικητικών ερευνών άρα χρειαζόμαστε την Όλαφ γι' αυτό υπάρχει η Όλαφ και υπάρχει η Όλαφ και διενεργεί έρευνε. Κάθε χρόνο κάνουμε έρευνε, Πέρσι σπάσαμε ρεκόρ, πάνω από 300 έρευνε κάναμε για αδικήματα, για εγκλήματα πιφ. Πέρσι συστήσαμε προς ανάκτηση περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ. Σε λίγες μέρες θα δημοσιεύσουμε την έκθεσή μας όπου θα δείτε. Θα δείτε ότι η συνεισφορά της Όλαφ σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά την ανάκτηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσης που παρανόμως εδαπανήθησαν λόγω απάτης είναι ένα τέταρτο από όλε τι ανακτήσεις που γίνονται σαν αποτέλεσμα των ποινικών ερευνών από όλε τις αρχές των κρατών μελών. Η Όλαφ με 200 ερευνητέ έκανε τη δουλειά του ενός τετάρτου ε, του συνόλου όλων των άλλων υπηρεσιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι κάτι και το μόνο που έχουμε προστατεύει τα οικονομικά έρευνα για εγκλήματα κάτω των οικονομικών συμφερόντων στην την Ευρώπη. Αν η ΕΠΟ μείνει έχει στην πρόταση του Συμβούλιο, έχω, τη χρειαζόμαστε, δεν θα υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει ένα κενό, υπάρχει ένας χώρος που δεν καλύπτεται από την ΕΠΟ. Εμείς δεν κινηθούμε στα χωράφια της ΕΠΟ, εκτός αν η ΕΠΟ μας ζητήσει να μπούμε για να τη στηρίξουμε. Τι αυτή η περίπτωση θα ε, λειτουργήσουμε ως υπηρέτε υπό την διεύθυνση της ΕΠΟ. Αλλά σε όλους τους τομείς και σε όλα τα κράτη-μέλη που θα είναι εκτός εντολής και αρμοδιότητες ΕΠΟ είμαστε εμείς εκεί. Υπάρχει ανάγκη. Δεν θέλετε την Όλαφ, θα χρειαστείτε κάτι άλλο δεν έχετε την Όλαφ για να καλύψετε το κενό. Διότι όπως σας είπα θα δημιουργεί το παράδοξο. Αν δημιουργούσαμε δηλαδή την ΕΠΟ και μετά σαν αποτέλεσμα αυτού κάποιοι τομείς πιφ δεν θα ελεγχονται ευρωπαικω ευρωπαϊκώς πορφή. Κάποια κράτη-μέλη δεν θα συμμετέχουν στην ΕΠΟ και θα κέρδιζαν διότι δεν, είχαν, δεν θα είχαν κανέναν έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως σήμερα. Λοιπόν, είναι απλό για μένα. Το να έχεις τέσσερις φορείς, Eurojust, Europol κλπ. κλπ. είναι κάτι δίσκαμπτο. δεν είναι και τόσο προβληματικό. Σήμερα έχουμε τρεις φορείς. Eurojust, Olaf και τα κρατημέλη. Αύριο η απόφαση του Συμβουλίου, αν ακολουθεί σε αυτή την κατεύθυνση, θα είναι να δημιουργηθεί τέταρτο φορέα. Δεν το διαλέξαμε εμεί αυτό. Θέλαμε η ΕΠΟ να είναι ο μοναδικό φορέα. Όμω, αν η εντολή μειώνεται, εγώ δεν βλέπω το πρόβλημα που υπάρχει να έχουμε τέσσερι φορέ. Τέλο πάντων, με κάθε σεβασμό, το Eurojust δεν θα έχει αρμοδιότητες για εγκλήματα πιφ. Για τα κράτη-μέλη όμως για τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στην ΕΠΟ. Όπου υπάρχει ΕΠΟ, υπάρχει ΕΠΟ. Σαν δικαστική αρχή, σαν διοκτική αρχή, σαν εισαγγελία. Για τα κάτι μέλη που δεν συμμετέχουν στην ΕΠΟ, το Eurojust θα είναι σημαντικότατο. Αλλά δεν είναι πρόβλημα να έχουμε τρεις ή τέσσερις φορείς. Το πρόβλημα είναι τι κάνει ποιος. πώς οι θεσμοί θα δημιουργήσουν την ΕΠΟ. Αν δημιουργηθεί ως έχει με περιορισμένες αρμοδιότητες, δεν είναι αποκλειστικός δικαστικός ερευνητικός φορέας, συμπληρωματικός φορέας είναι. Και έτσι αντί για τρεις έχετε τέσσερις. Εσείς το διαλέξατε. Αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα αν σκοτώσετε ονδήποτε άλλον φορέα για να απλουστευθεί το σύστημα για να μειωθούν οι φορείς. Τι ούτω τρόπος θα χάσετε και κατά πολύ θα χάσετε ευρωπαϊκά εργαλεία για τη διενέργεια ερευνών για εγκλήματα πύφη. Υπάρχει πλήρη συμπληρωματικότητα. Είναι κάπως άκομψο και δίσκαμπτο, αλλά όχι λόγω της υπάρξεως πολλών φορέων, αλλά λόγω του άκομψου χαρακτήρα, θα έλεγα, της, ε, του ορισμού των αρμοδιοτήτων της ΕΠΟ όχι της Όλαφ, της ΕΠΟ. Ευχαριστώ θερμά. Εάν δεν υπάρχει α, ερώτηση αυτή τη στιγμή, θα παρακαλέσω να περάσουμε στο τρίτο κομμάτι με την Παρμπαρα Ματέρα, Προεδρεύουσα. Ευχαριστώ τη Μισελ Κόνινγκς ευχαριστώ τον κύριο Κέσλερ για τις ομιλίες σας, για τις απαντήσεις, ερωτήσεις και παραδίδω την έδρα στη Βάρβαρα Ματέρα. Ξεκινήσουμε τι εργασίε του τρίτου πάνελ όσον αφορά την όλη αναθεώρηση στο δικαστικό τομέα. Καλώ ορίζω του εμπειρογνώμονε και του επόμενου ε, ομιλητέ. Ο κ. Ιβ Μποτ, Γενικό Διοικητή του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Χαιρετίζω τη δεύτερη ομιλητρία. Μαρία Χωσέ Μαρτίνε, Διευθύντρια τη Νομική Υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου Χαιρετίζω την κυρία Τερέζα Μπλανσέ, Διευθύντρια του Τμήματος Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και χαιρετίζω τον κύριο Γνάσιο Παντρώνε, συντονιστή για διεθνείς υποθέσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ιταλίας. Για εκείνους που έχουν παρασύργασεις από την αρχή ήταν ένα εντατικό και ενδιαφέρον απόγευμα για πολλούς από εμά ήταν και μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε τις αμφιβολίες που υπάρχουν σε αφορά αυτό το θέμα που είναι σημαντικό και ευαίσθητο αλλά μας επέτρεψε η συζήτηση να δούμε τους επόμενους μελλοντικού στόχους κυρίως σαν ευρωβουλευτές να είμαστε ακόμη πιο πεπισμένοι για τις μάχες που δίνουμε σε αυτό το πάνελ. Μιλάμε για την αναθεώρηση του δικαστικού αυτού θέματος, τομέα. Είναι πολύ σημαντικό για τη δημιουργία της ΕΠΟ, όπως ξέρουμε αντιπροσωπεύει ένα θέμα που είναι ανοιχτό, που άπτεται σημαντικών θεμάτων για το Κοινοβούλιο. Είμαι πεπισμένη ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εξαρτάται και από τελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου των αποφάσεων της, ε, όσον αφορά την αναθεώρηση αυτή τη δικαστική. Υπάρχουν διάφορες λύσεις αναλλακτικέ πώς να θεσμοθετηθεί αυτός ο μηχανισμός. Θα πρέπει να προβλέπουμε όμως τρία διαφορετικά ενδεχόμενα. Το πρώτο ενδεχόμενο όπου υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δεύτερο ενδεχόμενο, αντιθέτως τα εθνικά δικαστήρια θα έχουν το νομικό έλεγχο στον αφορά τις αποφάσεις και στο τέλος ένα μεικτό σύστημα που προβλέπει τον ρόλο των εθνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όμως δεν θέλω ε, να αναφερθώ σε αυτά που θα υποθούν στη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ιβ Μποτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, να πω, είναι κάτι που πρέπει να το πω, την προσωπική μου μονογνώμη θα εκφράσω. Και ίσως αυτά που θα πω πάντα μιλώντας από προσωπικό, θα θεωρήσετε ότι επηρεάζονται από τα προηγούμενα καθήκοντα που είχα ασκήσει. Ήμουν εισαγγελέα στη Γαλλία. Και παραλαμβάνω ότι ε, Δεσμεύομαι απόλυτα για όλα όσα θα σας πω προσωπικά. Η σημασία της δημιουργίας Ευρωπαϊκής αγγελία για την προστασία των πολιτών είναι πολύ σημαντική. Και είναι και ένα άκρος πολιτικά ευαίσθητο θέμα. Το, η ευαισθησία αυτού του θέματος προκύπτει από την αντιμετώπιση του ποινικού ε, δικαίου. Το ποινικό δίκαιο ξέρουμε ότι πάντοτε έχει ένα αποτέλεσμα ένταξης, όμως θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι εδώ και καιρό προσαρμόστηκε στην μεταξύ το έγκλημα. Ενσωματώθηκε, εντάχθηκε το έγκλημα. Άρα, είναι σαφές ότι η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής εισαγγελία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χαιρετήσουμε ως πραγματική πρόοδο και ως κάτι που έλειπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, διαβάζοντας το σχέδιο που μας κοινοποιήθηκε, διαπιστώνουμε ότι το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η αρχιτεκτονική είναι πολύπλοκη κατά τη. Είναι σαφές βέβαια ότι το άρθρο, το άρθρο συγγνώμη, 86 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το σύστημα που επιλέγει, επιλέγει δεν μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι πιο απλό και από την άλλη πλευρά εάν λάβουμε υπόψη τη φύση της αγγελίας και την αποστολή της, ίσως είναι εφικτό να χαράξουμε κάποιες γραμμές που μπορούν να οδηγήσουν σε μία, κάποια απλούστευση παρόλα αυτά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη φύση της αγγελίας. Νομίζουμε ότι από τη συνθήκη προκύπτει ότι θα πρέπει να θεωρείται ως ένα δικαστικό όργανο αφενός, αλλά και ένα ενσωματωμένο στο εθνικό ένομο σύστημα δικαστικό όργανο αφετέρου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι και μια υποχρεωτική συνέπεια που απορρέπει το ίδιο το άρθρο 86 που λέει ότι ε, είναι ένα ε, δικαστικό όργανο η εισαγγελία. Γιατί χρησιμοποιεί τον όρο παρκέ στα γαλλικά, εισαγγελία, που δεν είναι ουδέτερος όρος και στην τελευταία φράση του τρίτης παραγράφου του άρθρου 86 χρησιμοποιεί ε, την φράση άσκηση ε, δημόσιου λειτουργήματος εξερσίς δε fonction publique. Επίσης, αυτή η διπλή διαπίστωση, δηλαδή η δικαστική φύση αφενός, αλλά και η ένταξη της αγγελίας στο εθνικό ε, δικαστικό σύστημα, κατά την άποψή μας, πρέπει να καθοδηγήσει κατά κάποιο τρόπο νομίζουμε και να υπαγορεύσει αν θέλετε σε ένα βαθμό Τη κατευθυντήριες γραμμή για τον έλεγχο θα πρέπει να διενεργείται. Τελικά, επειδή θα πρέπει να δρά μέσω των εθνικών δικαιοδοσιών, στο κλασικό σύστημα μιας ποινική δίωξης, στο πλαίσιο των εθνικών ποινικών συστημάτων, γιατί θα έπρεπε να εφαρμοστεί ε, διαφορετικός κανόνας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνθήκη κάνει τη συγκεκριμένη επιλογή. Δηλαδή, το να γίνει κάτι εντελώ διαφορετικό από το κλασικό σύστημα λειτουργίας μιας εισαγγελίας ε, στο εθνικό σύστημα ήταν μια δυνατότητα, υπήρχε η επιλογή αυτή, ήταν ανοιχτή πόρτα αν θέλετε και θεωρούμε διαβεσβήτητο το γεγονός ότι την έκλεισε αυτή την πόρτα η συνθήκη. Και αφού την έκλεισε, ε, απλουστεύεται και το όλο θέμα, διότι τελικά σε τι χρησιμεύει η εισαγγελία, μια αρχή παρόμοια με μια εθνική αρχή. Στη δίωξη, στο να κάνει δίωξη, ε, ποινικέ διώξει. Ε, η απόφαση λοιπόν είναι μια απόφαση σε σχέση με το μου και την νομιμότητα που υπόκειται στην επιλαμβανόμενη δικαιοδοσία αν υπάρξει καταγγελία κάποιου περιστατικού από την όλα παραδείγματος χάρη, σε μια εθνική δικαιοδοτική αρχή, παρότι η ίδια η αρχή αυτής της καταγγελίας αμφισβητείται, το δικαστήριο λέει ότι δεν έχει αρμοδιότητα, γιατί η εθνική δικαιοδοτική αρχή που επιλαμβάνεται αυτής της καταγγελίας θα πρέπει να δώσει τη συνέχεια, τη δέουσα Άρα να εκτιμήσει το βάσιμο και την εγκυρότητα. Την νομιμότητα, συγγνώμη. Τώρα, αν μια απόφαση μεταφέρει την αρμοδιότητα αυτή από ε, την εισαγγελία στο δικαστήριο θα ήταν κάτι αντίθετο με το πνεύμα της συνθήκης. Άρα θα ήταν διαφορετικό το σύστημα, όχι αυτό το οποίο θέλει το άρθρο 86 πάντα μιλάμε για την πιστοποίηση του βάσιμου και της νομιμότητας. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την αποστολή τη διοκτική, θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε την εξή διαπίστωση. Η απόφαση για μία δίωξη, όπως λέει και η συνθήκη, αποσκοπεί και στη συλλογή πληροφοριών, την έρευνα, την ε, εκδίκαση μιας υπόθεσης ε, ε, και αυτή η απόφαση περί δίωξης θεωρούμε ότι ναι μεν πρέπει να συνεπάγεται τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Υπάρχει η δικαστική και αστυνομική συνεργασία. Οι διατάξεις λοιπόν του κανονισμού πιστεύω ότι θα μπορούσαν να επαρκούν ώστε το πραγματικό πρόβλημα τη εφαρμογή να μην τίθεται καν. Διότι καταλαβαίνω πολύ καλά ότι η λειτουργία μια αγγελική αρχής μπορεί να φαίνεται κάπως μυστηριώδη, σε ε, ε, απριόρι, υπάρχουν συστήματα στα κράτη-μέλη, ε, τα 28 που έχουν καθημερινή επικοινωνία και όταν μπορούν και όσο μπορούν να δρούν σε συντονισμό μεταξύ τους, όπως γίνεται μέχρι στιγμής υπό την Eurojust. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να διευκολύνουμε την κατανόηση όλων αυτών, ε, αν μου μία υπόδειξη στο κείμενο που αποσκόπησε τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δικαιοδοσιών. Μήπως θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε αυτήν την έκφραση νόγμα μινιμάλ, κατώτατα πρότυπα. Είναι αρνητική η χρειά που έχει και θα έπρεπε να αντικατασταθεί από το ε, «garantie εντεγοζάμπλ συζητήσιμη εγγύηση, Μπορεί αυτό να συγκεκριμενοποιηθεί σε εθνικό δίκαιο, αλλά αν δεν γίνει αυτό θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας. Αυτά τα κατώτατα πρότυπα, κατώτατοι κανόνες, θέλω να μας πούν ουσιαστικά εμέσως ότι δεν είναι καλής ποιότητας ε, ο κανόνας. Δεν ισχύει όμως σε καμία περίπτωση αυτό. Γι' αυτό και λέω ε, ότι με αυτή την υπόδειξη που σας κάνω πιστεύω θα διευκρινιστούν κάποια πράγματα και θα αποφευθούν και πολλές δυσκολίες. Γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του και όπως πρέπει. Ένα άλλο παράδειγμα. Απόφαση για μη δίωξη. Σας είπα τι πιστεύω για την απόφαση για δίωξη, που ένα από το πω είπα στην κρίση της δικαιοδοτική αρχή Τώρα, απόφαση για μη δίωξη. Ταξινόμηση αμπινίσιο. Πού έχουμε πρόβλημα εδώ, αφού υπάρχει αρμοδιότητα συντρέχουσα. Mm. Αμέσως ξεκινά ε, η δυνατό, αρχίζει η δυνατότητα για ένα, ε, μια εθνική δικαστική αρχή να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, αν το κρίνει απαραίτητο. Η επιλογή της δικαιοδοσίας, που θα πρέπει να γίνει η συγκέντρωση, γιατί εξορισμού σε δυσυνοριακό επίπεδο, σε δυσυνοριακό τομέα. Η δικαιοδοσία που επιλέγεται όμως είναι η δικαιοδοσία που είναι εθνική δικαιοδοσία και λειτουργήμα του Εθνικού Δικαστή είναι να αξιολογεί την ίδια την αρμοδιότητα. Αλλά αν υπάρχει μια αμφιβολία, και μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα από αυτή τη συγκέντρωση, απόρρια του κανονισμού που εγκαθιδρύει την την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχει και η δυνατότητα ε, υποβολής προδικαστικού ερωτήματος προς το δικαστήριο. Και το ξέρουμε, είναι καθημερινό φαινόμενο να υποβάλλονται τέτοια ερωτήματα. Έχω ακούσει για διάφορα συστήματα και όλα αυτά τα συστήματα, λυπούμε που έχω ξεπεράσει λίγο το χρόνο που είχα αρχικά στη διάθεσή μου, αλλά δεν πρέπει να μου δίνετε το λόγο να μιλήσω για την εισαγγελία, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να μην σταματάω. Λοιπόν, ναι, πώς να σας το πω λοιπόν, ε, ένα τέτοιο σύστημα, ένα άλλο σύστημα έχει μια διπλή δυσκολία. Μιλήσαμε για τις διαφορές της δικαστικές, διενέξεις. Τι θα γίνει. Ε, έχουμε μια σχέση εδώ, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Εθνικές Εισαγγελίες. Και η εισαγγελία δεν είναι το κράτο, ε, είναι η δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη. Και το καθεστώ που προβλέπεται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσε να ε, εξυπηρετήσει και ένα, να υπηρετήσει ω ένα εθνικό μοντέλο για την αντίστοιχη Εθνική Εισαγγελία. Είμαστε σε ένα ε, σύστημα διαφορετικών αναλύσεων κτλ. και ερμηνεών. Έχουμε την Εθνική Εισαγγελία από τη μία, όπου ένα μέλο συγκεκριμένο Έχουμε τον εντεταλμένο ε, Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα που εντάσσεται στο εθνικό σύστημα που έρχεται σε αντίθεση και σύγκρουση με την αρχή, την ίδια. Τον προϊστάμενό, αν θέλετε. Άρα, από ανθρώπινη, πώς να το πω, πλευρά, θα πρέπει να μπορούν να συμβιώνουν αυτοί. Πρέπει να είναι δυνατόν να ε, επικοινωνούν, να συνεννοούνται. Και σίγουρα αυτή τη φορά, αν δούμε και το θέμα της εθνικής κυριαρχίας, ε, υπό αυτή την έννοια θα ανοίξουμε την πόρτα για πολιτική ε, έποψη, πολιτική αντιμετώπιση του ζητήματος που δεν έχει να κάνει όμως με πολιτική αλλά με δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω πάσο ότι σε περίπτωση αμφιβολία υπάρχει η δυνατότητα υποβολή προδικαστικού ερωτήματο. Και εκεί ξέρουμε τι κάνει η δικαιοσύνη. Ή θα παραμείνει και θα έχει το ρόλο αυτό, ή αλλιώ πρέπει να αλλάξουμε και τη σύνθεση του δικαστηρίου και να δημιουργήσουμε ένα ειδικό σώμα. Γιατί, για να ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο, μα δεν θέλει να ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο το δικαστήριο. Αρνείται να το κάνει. Αυτά, σταματώ εδώ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα απλά να σας εκφράσω το βάθος της σκέψης μου. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι καλή ιδέα, επαναλαμβάνω, πρέπει να γεννηθεί, αλλά ας του επιτρέψουμε και να ζήσει ως όργανο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπότ. Ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο να σας ακούω. Σας υπόσχομαι θα σας καλέσουμε και στο μέλλον και τους εμπειρογνώμονες που έχουμε σήμερα στα τρία πάνελ, διότι δυστυχώς ο χρόνος στη διάθεσή μας εδώ στο Κοινοβούλιο είναι πάντα πολύ περιορισμένος εντός των επιτροπών. Αλλά δεσμευόμεθα ούτως ώστε να υπάρξουν άλλες συναντήσεις επ' αυτών των θεμάτων και των θεμάτων του δικαστηρίου. Τώρα όμως θα περάσω το λόγο στην κυρία Μαρία Χωζέ Μαρτίνε, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην αρχή αυτή τη νομοθετική διαδικασία, το Δεκέμβριο του 2014, για να θυμάται, η νομική υπηρεσία εκλήθηκε να δώσει γνωμοδότηση για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εισαγγελία και ιδιαίτερα το άρθρο 36 της πρότασης κανονισμού και ιδιαίτερα η Επιτροπή σας ζήτησε εάν σημαίνει το άρθρο αυτό πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα είναι σε θέση να αξιολογήσει εάν πράξεις της ΕΠΟ είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και επιπλέον εάν αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με το άρθρο 263 για την αναθεώρηση νομιμότητας και το 267 για τις προδικαστικές αποφάσεις. Η απάντηση νομικής υπηρεσίας ήταν απερίφραστη. πράξη η παράληψη του Ευρωπαίου Εισαγγελέα χαρακτηριζόμενη ως αντίστοιχη εθνικού εισαγγελέα δεν επιτρέπει την προσφυγή το 263 και 267 για πράξη παραλήψης ή παραβίαση παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, αυτό άμεσα απευθείας δηλαδή παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και βέβαια και την αναλογικότητα με τη δυνατότητα της αποκατάστασης που προβλέπει το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, το άρθρο 36 της προτάσεως κανονισμού εγείρει σοβαρές ανησυχίες προς την ομιμότητά του. Όσο σαφής και να είναι η απάντησή μας αυτή, βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μια υβριδική μορφή ε, χήμερα μεταξύ του ε, εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν μπορεί να είναι ποτέ απλή δηλαδή μια απάντηση. Το άρθρο 36 παράγραφος 1 θα μπορούσε να αποκλείει την διεκδίκηση δικαιωμάτων ε, διαδίκου έναντι δικαστηρίων κρατών μελών. Αυτό βέβαια δεν καταργεί τα ένδικα μέσα τα ίδια, αλλά η άσκηση και η ε, επίτευξή τους θα εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο. Με το νομικό πλάσμα δε, δυνάμει το οποίο θεωρείται εθνική αρχή ΕΠΟ, δίδεται αρμοδιότητα στα εθνικά δικαστήρια να κρίνουν ζητήματα νομιμότητας δράσεως ευρωπαϊκού οργάνου. Παράλληλα, στο ίδιο άρθρο, η δεύτερη παράγραφος ορίζει ότι η διατάξη του εθνικού δικαίου μόνο και μόνο επειδή παραπέμπει σε αυτά ο κανονισμός, σε αυτές ο κανονισμός, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως καλύπτουσες τις προϋποθέσεις για την προδικαστική εξέταση. Η διάταξη αυτή λοιπόν, 36.2, διαβαζόμενη σε συνδυασμό με το υπαριθμό 1 συνεπάγεται πως δεν μπορεί το δικαστήριο να εξετάσει την νομιμότητα ούτε καν σε προδικαστικό επίπεδο των πράξεων του Ευρωπαίου Σαγγελέα. Με βάση το χάρτη και τα άρθρα της συνθήκης λοιπόν έχουμε πρόβλημα προς την άσκηση των ανδίκων μέσων. Στο χάρτη των δικαιωμάτων καταγράφεται η απέτηση για την δυνατότητα αποκατάστασης δικαιωμάτων σε περίπτωση παραβιάσεως των δικαιωμάτων και ελευθεριών που εγγυάται το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, δυνάμει του άρθρου 51 του χάρτη και έχει ιεραρχική σχέση ανώτερη ως προς τις λοιπές ευρωπαϊκές διατάξεις. Δεν είναι απόλυτο το δικαίωμα σε ένδικα μέσα. Μπορεί να υπαχθεί σε δικαιολογημένος όμως δυνάμει του άρθρου 52 του χάρτη περιορισμού, σε δικαιολογημένους ε, περιορισμούς με βάση την αρχή και της αναλογικότητας. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος και πάνω απ' όλο κατάλογος των ε, φορέων και οργάνων στα οποία ισχύει είναι δεσμευτικός και περιοριστικός και άρα δεν μπορεί να διευρυνθεί. Είναι αυτά που καταγράφει το άρθρο 57. Δεν μπορεί να τροποποιηθεί αυτός ο κατάλογος από ένα νομοθετικό όργανο. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει πως ο ορισμός του κατά πόσον ένα σώμα είναι σώμα ή φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνιστά διακριτική ευχέρεια των ε, νομοθετών. Βλέπετε επίση μια σειρά από 11 μέσα για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και την νομιμότητα στην Ένωση, καλύπτοντα έτσι ε, με διαδικασία δικαστική στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και τις υπηρεσίες και σε σχέση με το δευτερογενές δίκαιο και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα για την αφισβήτηση πράξεων των οργάνων της Ένωσης, των παραλήψεων αυτών και βέβαια ε, προσφυγή για την αποκατάσταση δικαιωμάτων η αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης από νομοθετήματα και αποφάσεις πράξης ή παραλήψεις των ευρωπαϊκών οργάνων. Η συνθήκη θεσπίζει λοιπόν ένα πλήρες σύστημα ένδικων μέσων που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εξετάσει την νομιμότητα των μέσων των αποφάσεων που οθετούν τα, θεσμικά, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μόνο με τροποποίηση των συνθητών μπορεί να αλλάξει. Δεύτερο γενές, το παράγωγο λεγόμενο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υποκαταστήσει και να τροποποιήσει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπως αυτές απορρέουν από τη συνθήκη. Και αυτό αφορά όχι μόνο άμεσες πράξεις ή δράσεις αλλά και προδικαστικές αποφάσεις για το πρωτογενές και την ερμηνεία του πρωτογενού και παράγωγου δικαίου και των νομοθετημάτων λοιπόν πράξεων. Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να αξιολογήσει την τήρηση του νομικού του ένομου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω των προδικαστικών αποφάσεων. Το διφυλονικούμενο ζήτημα είναι εάν το άρθρο 86 της νομικής βάσης επιτρέπει εξαιρέσεις στο καθεστώς αυτού. Η δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πιστεύουμε ότι ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία παρά τις ιδιαιτερότητες της δυνάμει του άρθρου 86 και ιδιαίτερα σε σχέση με το ρόλο που διαδραματίζουν αυτές οι διατάξεις τα εθνικά δικαστήρια. Η δεύτερη παραγραφός του άρθρου 86 ε, καταρχάς αναφέρεται σε δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων. Αυτό όμως έχει να κάνει μόνο με την εισαγγελική λειτουργία και όχι με την διερεύνηση. Η εισαγγελική λειτουργία της εφαρμογή άπαξ και η εισαγγελική αρχή έχει επαρκή στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή έχει επαρκή στοιχεία για να ε, προσαγάγει σε δίκη ε, και να προβάλλει αποδεκτικά κτλ. Αλλά αυτό δεν αλλάζει του δικαιοδοτικούς κανόνες που ισχύουν εν γέννη για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επίσης η τρίτη παράγραφος του άρθρου 86 που ορίζει πω υπάρχει υποχρέωση για συμπερίληψη στον κανονισμό ο οποίος θα ορίζει τους κανόνες για, δικαστική, ε, για το δικαστικό έλεγχο πράξεων ή παραλήψεων κατά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής ε, δεν λέει τίποτε συγκεκριμένο ως προς τη δικαιοδοσία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ωστόσο, ε, εξαίρεση από την ε, αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα είχε πολύ σημαντικές συνέπειες για την δικαιοδοσία. Δηλαδή θα πηγαίναμε στο άρθρο 270 που αποκλεί ε, τις αστυνομικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές ε, από, τη δικαστική, το δικαστικό έλεγχο ή άλλο τομέα όπως αυτό της ε, εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας. Δεν αναφέρει λοιπόν το άρθρο 86, δεν αναφέρεται το άρθρο 86 ως ε, άρθρο το γενεσιουργό ή ασδήποτε ε, εξαίρεσης εν προκειμένου. Και η τρίτη παράγραφος του 36 πρέπει να αναγνωστεί και να γίνει κατανοητή με βάση το θεμελιώδες δικαίωμα στην ε, άσκηση και αποκατάσταση με ένδικα μέσα. Άρα πρέπει να έχει μάλλον διασταλτική παρά συσταλτική ερμηνεία και αυτό θα πρέπει ε, να έχει σαν αποτέλεσμα μια αποτελεσματική άσκηση ενδίκων μέσων και υποκατάσταση δικαιωμάτων. Για μας λοιπόν το άρθρο 86 παραγραφός 3 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαιοδοσία και να περιορίσει τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία ουσιαστικά ορίζεται το άρθρο 19 της Ενδείξης τη Λειτουργία και τα άρθρα 260 κλπ και επόμενα τη Σύνθήξη τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό καλύπτει και τις πράξεις αλλά και τις παραλήψεις του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αυτή είναι η αρχική μας λοιπόν ανάλυση. Οι ε, διατάξεις στην προτινόμενη στο νομοθέτημα, νομοθέτημα γύρουν πολύ σοβαρά ε, ερωτηματικά σχέση με την νομιμότητά του. Πάντως δεν ισχύουν για πράξεις ή παραλήψεις του Ευρωπαίου Εισαγγελέα που μπορούν να εγγραφούν στην εισαγγελική λειτουργία πριν από την παραπομπή σε εθνικά δικαστήρια, καθώς δεν προβλέπεται δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διαφυλαχθούν αυτές οι αρμοδιότητες για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όποιος ισχυρίζεται ότι μόνο τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να έχουν ε, δικαιοδοσία, ε, ε, προφανώς εννοεί ότι αυτή προκύπτει άπαξ και ασκηθεί η ποινική δίωξη. Και βέβαια τα κενά στην δικαιοδοσία θα πρέπει να καλούνται από κοινού μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Δικαστηρίων για να υπάρχει μια ουσιαστική απόδοση δικαιοσύνης. Η Προεδρία του Συμβουλίου στο τελευταίο έγγραφο της 22ης ε, Δεκεμβρίου του 2015 είχε σημειώσει μια διαφορετική εκδοχή του άρθρου 36, όπου η δεύτερη παράγραφος αποκαθιστά τη δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής, έκδοσης προδικαστικής απόφασης και άρα είναι σύμφωνη από ό,τι βλέπουμε με τη δική μας ανάλυση. Από την άλλη όμως έχουμε τις αμφιβολίες μας για την προτινόμενη πρώτη παράγραφο, όπως την προτείνει η Προεδρία. Ναι, ναι, ό, τελειώνω, τελειώνω. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν αυτή είναι μια τελική εκδοχή. Πάντως... Οι ερευνητικές ε, δραστηριότητες δεν μπορούν να αποκλειστούν με μια τέτοια διάταξη. Και πάντως, εάν τροποποιούν την, ε, τις ένομες σχέσεις του εμπλεκομένου διαδίκου, και τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου δεν μπορεί να ισχύουν. Μια μερική, ένας μερικός αποκλεισμός του άρθρου 36 θα πρέπει να προχωρήσει με μια πιο σαφή ε, περιγραφή για να μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική ανάλυση. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ Τερέζα Μαρτίνες. Δεν μ' αρέσει που σας διακόπτω, αλλά δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τερέζ Μπλανσί Διευθύντρια του Τμήματος Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα εκφραστώ προσωπικά. Είμαι διευθύντρια τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, αλλά βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, μπορώ να εκφραστώ τον ονόματι του Συμβουλίου, τον ονόμα τη νομική υπηρεσία, διότι οι εργασίε ε, εξελίσσονται, δεν έχει ολοκληρωθεί πλέον η εργασία, είναι περίπλοκο θέμα Ήδη εδώ και τρία χρόνια διαρκεί και παραπάνω η συνθήκη δημιούργησε λοιπόν δύο υβρίδια θα λέγαμε. Ένα υβρίδιο που είναι γνωστό, είπατε εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, την κοινή και την ασφάλεια είναι ένα υβρίδιο μεταξύ δύο θεσμών και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μάλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει και άλλη ε, αρμοδιότητα. Το δεύτερο υβρίδιο είναι αυτό που συζητούμε σήμερα, που είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο, που είναι ένα υβρίδιο που συμπεριλαμβάνει έναν φορέα ευρωπαϊκό και έχει μια λειτουργία και ρόλο ε, εντός των εθνικών θεσμικών φορέων. Είναι ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που καλείται να κινηθεί εντός των ε, εθνικών δικαιοδοσιών κατά των παραβάσεων ΠΙΦ. Ε, λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο Συμβούλιο και αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ο έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων αυτής της αγγελία που είναι ένα όργανο της Ενώσεως που συνήθως το δικαστήριο ελέγχεται στο άρθρο 263 και το 267 όσον αφορά τον έλεγχο των παιδικαστικών θεμάτων και την ερμηνεία αυτών προβλέπει ότι το δικαστήριο είναι αρμόδιο επίση και για τα όργανα και του οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, όχι μόνο για τα θεσμικά όργανα. Το λεξιλόγιο αυτό ολοκληρώθηκε και από τη συνθήκη της Λισαβόνα τότε. Λοιπόν, το θέμα που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό το άρθρο 86 παράγραφος 3 που δίνει τη δυνατότητα στον νομοθέτη να καθορίσει τον κανονισμό, τους κανόνες για τον έλεγχο, των νομοθετικό όσον αφορά τις διαδικασίες που θετεί σε ε, τη εκτελέση των καθηκόντων του, σε ποιο βαθμό το άρθρο αυτό επιτρέπει να είναι μια, είναι μια νομική βάση που δίνει τη δυνατότητα στον νομοθέτη να παρεκκλίνει από τους κανόνες και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όπως τα γνωρίζετε, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου του 2013 έναντι της περιπλοκότητα του βριβίου προσπάθησε να προβεί σε μια απλούστευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε και ο Γενικός εισαγγελέα, να περιοριστούν οι αρμοδιότητες του δικαστηρίου μόνο όσον αφορά, αφορά την ερμηνεία και την εξέταση προδικαστικών θεμάτων και των θεμάτων που αφορούν την ισχύ, αυτά που καλύπτει ο κανονισμός και αρμοδιότητα που έχει όσον αφορά τι μη συμβατικέ συμβατικές ε, του δικαστηρίου, δηλαδή άρθρο 3 και 5 του 69. Αποκλείεται η αρμοδιότητα του δικαστηρίου από όλα τα άλλα. Δηλαδή τα δικονομικά μέσα, τι διαδικασίες που ακολουθεί βάση της παραγράφου 1 το 36.1 και το 36, άρθρο 36 αφορά τις εξαιρέσεις βάσει ε, μια, μιας διπλού καθορισμού. Άρθρο 36 παράγραφος 1 προσωμιώνει με εθνική αρχή το, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για όλα τα ε, δικονομικά. Υπάρχει ο έλεγχος άμεσος και έμεσος ε, από πλευράς δικαστηρίου για την ακύρωση και έμεσα μέσω της, παρα, της της προδικαστικής όλα, τα, όλα εκφεύγουν τα δικονομικά ε, από την, ε, το δικαστήριο τεχνικό και κυρίως αυτές που βασίζονται στον κανονισμό. Αυτή είναι η συνέπεια της παραγράφου 1 όπως ε, προτάθηκε τότε. Η παράγραφος 2 λοιπόν το άρθρο 36 καθορίζει με άλλο ενδεχόμενο νομικό. Δηλαδή καθορίζει ότι οι εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται από τον κανονισμό δεν θεωρούνται ότι αφορούν δίκαιο της ενώσεως για τον προδικαστικό έλεγχο. Αυτό καταλήγει στο να εξαιρεθούν από, τις εθνικές από την ερμηνεία την προδικαστική, αυτό εξαιρεθεί στην αιτιολογική σκέψη 39, και όταν οι εθνικές διατάξεις εφαρμόζουν το δίκαιο της ενώσεως, δηλαδή την οδηγία PIF ή την οδηγία που αφορά την ενορμόνιση των ποινικών διαδικασιών. Συνεπώ, προφανώ, όσοι συζητήσει στο Συμβούλιο, ένα από τα πρώτα ερωτήματα που ετέθη ήταν το εξή. Ποιο ήταν το εύρο των εξουσιών παρεκκλήσεω ε, του νομοθέτου από το άρθρο 86 ε, παράγραφος 3. Όπω έλεγε η συνάδελφο Μαρία Χωζέ, όταν συγκρίνουμε το 86-3 με τι άλλε διατάξει των συνθήκων που παρεκλείουν, δίνουν παρεκκλήσει από του δικαστηρίου, βλέπουμε ότι υπάρχουν φορέ στον αφορά το άρθρο 74 παράγραφος 9, 108 ή 348 δεύτερο, δεύτερη παράγραφο που καθορίζει τις παρεκκλήσεις λέει κατά παρέκκληση από τα άρθρα κλπ. Λέει διατύπωση. Όσον αφορά τη δυνατότητα που δίνεται στο νομοθέτη τη ενό στο άθρο 263 πέμπτη παράγραφος να προβλέπει στις πράξεις που δημιουργούν οργανισμούς μια δυνατότητα ιδιαίτερη όσον αφορά την ακύρωση αποφάσεων, αυτό το άρθρο δεν δίνει δυνατό στο νομοθέτη να παρεκκλίνει πλήρω από τι αρμοδιότητε του δικαστηρίου όσον αφορά τη δράση ακύρωση αποφάσεων. Αυτά είναι μόνο παραδείγματα. Λοιπόν, το θέμα που τίθεται είναι κατά πόσο η διατύπωση χρησιμοποιείται στο άρθρο 86 που επιτρέπει τον καθορισμό κανόνων για τον έλεγχο των διαδικασιών του εισαγγελία εξαιρεί το δικαστήριο που άμεσο ή έμεσο έλεγχο των διαφόρων δικονομικών κινήσεων του, της αγγελίας. Ξέρουμε ότι στην ομολογία την κλασική του δικαστηρίου εφόσον είναι, κάτω, είναι ένωση δικαίου η ένωση λέει ένα πλήρες σύνολο δυνατοτήτων διαδικασιών για να μπορούν να ελέγχουν την ομότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων προβλέπει ότι μείωση περιορισμοί της πρόσβασης στην προσφυγή για ακύρωση αντισταθμίζεται από την πρόσβαση στην προδικαστική ιδίωδο έγκρισης όπως γνωρίζετε και όπως διαπιστώνεται και από το κείμενο που προτέθηκε στην αρχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα προδικαστικά και την ερμηνεία σε κάποιες περιπτώσεις αλλά όσον αφορά και την ισχύ αυτά ξερούνται από το κείμενο. Λοιπόν, ένα, ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβε το Συμβούλιο για αυτή την περίπτωση ήταν να διαγράψει την παράγραφο 2 του άρθρου 36 διότι έξερε την προδικαστική πρόσβαση ε, όσον αφορά την ερμηνεία των εθνικών διατάξεων που καθίστανται εφαρμοστέ από τον κανονισμό. Δηλαδή, όπω έλεγα προηγουμένω, οι εθνικέ διατάξει που εφαρμόζουν το δίκαιο τη ενώσεω, παραδείγματο χάρη την οδηγία ΠΙΦ την ίδια ή την οδηγία εναρμονίσεω στον τομέα των ποινικών διαδικασιών, βεβαίω αυτό δεν έπρεπε να εξαιρούνται από την ε, δικαιοδοσία να ερμηνεύει το δικαστήριο. Απεκαταστάθη η δυνατότητα του δικαστηρίου λοιπόν στη διατύπωση του εναρμονή Συμβούλιο. Έμενε το θέμα του ελέγχου τη νομιμότητα των ποινικων διαδικασιων βεβαιω αυτο δεν επρεπε να εξαρτούνται απο την δικαιοδοσια να ερμηνευει το δικαστηριο απεκατασταθη δυνατοτητα του δικαστηριου λοιπον στη διατυπωση του κειμενου που προεβλεψε το συμβουλιο εμενε το θεμα του ελεγχου τη νομιμοτητα των διαδικαστικών της εισαγγελία. Και εκεί η λογική ποια ήταν, να κάνουμε διάκριση δύο φάσεις. Πρώτα είχαμε τη φάση πριν να επιληφθεί η εθνική νομοθεσία και δεύτερον μετά και να εξεταστούν εν συνεχεία τα θέματα από την πλευρά της άμεσης πρόσβασης για την ακύρωση και τον έλεγχο του προδικαστικό για την ισχύ των αποφασών αφορά την έμεση προσέγγιση. Ο έμεσος έλεγχος για τα προδικαστικά ζητήματα, κυρίως για, για όσα έχουν αποφασιστεί πριν από... να επιληφθεί η δικαιοδοσία, δεν μπορούσαν να αποκριστούν. Λοιπόν, η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε, ούτω ώστε να εφαρμόσετε το άθρο 267 των συνθήκων για τουλάχιστον για αυτά τα θέματα. Όσον αφορά την άμεση προσέγγιση, αρμοδιότητα για ακύρωση, δύο στιγμές εξετάζονται μετά την επίληψη της δικαιοδοσίας ή πριν. Πριν επιληφθεί η εθνική δικαιοδοσία. Όπως λέει η συνθήκη, από τη στιγμή που ασκεί δημόσια δράση ενόψεων των δικαιοδοσιών ή εισαγγελία, προσωμιάζει σε εθνική αρχή και ο έλεγχος ακολουθεί. Αυτή είναι η ερμηνεία των συνθήκων και αυτό είπε προηγουμένως ο κύριος Μπότ. Όσον αφορά την φάση που προηγείται της επιλήψεως της δικαιοδοσίας, η εισαγγελία δεν μπορεί να προσωμιωθεί σε μια εθνική αρχή όσον αφορά όλα όσα εγκρίνει πριν επιληφθεί η δικαιοδοσία. Το κριτήριο το λογικό που ακολουθείται είναι το εξή. Ποιο δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόσει η εισαγγελία. Η εισαγγελία εφαρμόζει βασικά το εθνικό δίκαιο ή αυτό τη ενώσεω, τον κανονισμό με άλλα λόγια. Αν η εισαγγελία εφαρμόζει βασικά το εθνικό δίκαιο, λοιπόν το να προσωπηθεί με εθνική αρχή, αποκλείοντα έτσι την αρμοδιότητα του δικαστηρίου, είναι κάτι αποδεκτό απολύτως. Παραδείγματο όσον αφορά τα μέτρα ερευνητικά που εντέλει η εισαγγελία πριν επιληφθεί η εθνική δικαιοσία και εκτελούνται από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα. Είναι λογικό λοιπόν ότι ο δικαστικός έλεγχος αυτών των μέτρων των ερευνητικών θα πρέπει να αναλαμβάνεται από τις εθνικές αρχές. Αν όμως η εισαγγελία εφαρμόζει ουσιαστικά τον κανονισμό η άμεση αρμοδιότητα του δικαστηρίου για να ελέγχει την νομιμότητα των πράξεων τη αγγελία που υπαθυμίζουν ένα όργανο τη ενώσεω θα πρέπει να διατηρηθεί. Και ο τρόπο κάποιε πράξει διαδικαστικέ που υιοθετεί άμεσα η εισαγγελία εν εφαρμογή του κανονισμού, όπω η πράξη μα των οποίων δηλώνει αρμοδιότητα, επιλεγεί τη αρμόδια δικαιοδοσία εδαφικά ε, και, διά, και διάφορα άλλε ρυθμίσει, εφαρμόζει δηλαδή η εισαγγελία, τον κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ή γίνεται κάποια συναλλαγή. Όταν όλα ρυθμίζονται μέσω του κανονισμού και εφαρμόζεται ο κανονισμό, και η προσφυγή σε ακύρωση θα πρέπει να μπορεί να ανοιχθεί. Είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζεται, εν κατακλείδη, όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται στο Συμβούλιο και τις συνεισφορές που έγιναν για τη νομική ανάλυση, οι δυνατότητε εθνικέ δικαιοδοσίε να κάνουν παραπομπέ προδικαστικέ όσον αφορά την ερμηνεία δεν θα πρέπει να περιορίζονται και δεν γίνεται κάτι τέτοιο και κάποιε δικαστικέ δικονομικέ πράξει πριν επιληφθεί η δικαιοδοσία και που βασίζονται άμεσα επί του κανονισμού σε επιλογή ε, ε, του που γίνεται, ποιο είναι υπεύθυνο ε, και οι διαδικασίε ενώπιν των δικαστηρίων ε, όπως κατεπίγουσες προσφυγές. Αυτά βάση του, ε, ρυθμίζονται βάσει του άρθρου 263. Ε, Σας ευχαριστώ κυρία Μπλαμσέτ και εμείς ελπίζουμε ότι αυτό το υβρίδιο που δημιουργήθηκε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπορεί τελικά να μορφοποιηθεί μετά από χρόνια όπου να δημιουργηθεί, να γεννηθεί, να αποκτήσει σώμα, να μεγαλώσει, να περπατήσει από μόνο του, να σταθεί στα πόδια του. Λοιπόν, κλείνοντας τις εργασίες, καλώ τον κύριο Πατρόνε που είναι συντονιστής για τις διεθνείς υποθέσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ε, Ιταλίας που παρακολούθησε από πολύ κοντά τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας να πάρει το λόγο. και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είμαι ο τελευταίος, ύστερα από μια συζήτηση πλούσια σε προτάσεις και συστάσεις. Και είμαι βέβαιος ότι θα χαρείτε αν περιορίσω σε λίγο χρόνο την ομιλία μου. Θα περάσω πολύ γρήγορα στα σημεία τα οποία θεωρώ ακόμα διαφλονικούμενα. Το άρθρο 36, το σχέδιο της Επιτροπής, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί το ζήτημα της δικαστικής επισκόπησης προκύπτει ήδη κατά τη φάση επεξεργασίας του εγγραφού, του σχεδίου και πρέπει να δούμε εάν έναντι αυτού του σχεδίου για τη σύσταση αυτού πρώτου οργάνου δικαιοσύνης ευρωπαϊκής και άρα θα πρέπει και άρα εκείνου που θα πρέπει να τηρεί τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργίας της και άρα του ομοσπονδιακού πλέγματος θα λέγαμε μπορεί να υπάρχουν αρμοδιότητες για κάποιον δικαστή περί επαλήθευσης κάποιων νομοθετημάτων Ήδη από το 2009-10 είχαμε κάποιες αμφισβητήσεις και συζητήσεις για το θέμα αυτό με μια πρώτη ιδέα ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια ποινική δικαιοσύνη, ένα ποινικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πολύ αξιόλογους δικαστές του Λουξεμβούργου. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ζήτημα που προκύπτει. Τι είδους αρμοδιότητες μπορεί να έχει ο δικαστής του Λουξεμβούργου και τι αρμοδιότητες θα αναλάβει ο Ανδαλούσιος ή ένας από τις βαλτικές χώρες δικαστής, ο εθνικός δικαστής του ΣΥΠΗΝ, ε, με βάση τις εθνικά συστήματα δικαιοδοσίας. Και δεν είναι απλή απάντηση, γιατί στη συζήτηση αυτή τίνουμε πάντα και πρέπει εδώ να διορθώσω, αν μου επιτρέπετε, την ε, Πρόεδρο. Είμαι αντισαγγελέα στο το Δικαστήριο Εισαγγελέα λοιπόν και άθελά μου πρωταγωνιστής του ποινικού δικαίου. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε κάθε θεσμός που ιδρύεται να έχει τη μέγιστη ε, αποτελεσματικότητα και κάθε εγγύηση απαραίτητη ε, για την προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε δηλαδή αυτό το στόχο που έχει η δικαιοσύνη να υπηρετήσει βεβαίως στην κοινωνία αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί και να στρεβλώνει τη θέση του κατηγορούμενου ε, και να τον θέτει σε δυσκολότερη μοίρα. Και θέλω για να εξηγήσω το εξής. Να πω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ε, να αναγνωριστεί ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων του δικαστή της Ένωσης, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Πρωτοβάθμιο ή Γενικό Δικαστήριο όπως τώρα λέγεται, αλλά αυτό είναι ένας άλλος προβληματισμός. Πάντως ε, κεντρικό χώρο δηλαδή ε, να αναγνωρίσουμε στο δικαστικό έλεγχο των ευρωπαϊκών ε, οργανών. αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να πάει για την υπερασπιση του μέχρι το Λουξεμβούργο, πράγμα το οποίο δεν είναι πλή υπόθεση, κοστίζει αρκετά και πάντως σημαίνει διάταξη ε, και διάθεση πόρων που δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν καταγράφηκε αυτό θένα, μόνο σε κάποιο κείμενο είχε αναφερθεί σαν υπόθεση, αλλά πάντως δεν προχώρησε. Και κάποιος ανέφερε νωρίτερα στη συζήτηση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση του 2013 ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή το πλάσμα δικαίου εκείνο βάσει του οποίου όλες οι πράξεις θα θεωρούνταν ως εθνικού χαρακτήρα, δηλαδή θα υπάγονταν στον έλεγχο του εθνικού δικαστή. Και έναντι και των συζητήσεων που ανέφερε και ο Γενικός Εγγελέας Μπού νωρίτερα, και για τον οποίο βέβαια τρέφω μέγιστο σεβασμό και τη δεσμερίζομαι απολύτως στις θέσεις του, αυτό σημαίνει ότι κάθε δικαστής της Ένωσης θα έχει τη δυνατότητα της δικαστικού ελέγχου για ασδήποτε απόφαση ε, του εισαγγελική Αρχής σε σχέση με την απόφαση, με κάποια απόφαση σχετική με τον κανονισμό και άρα κάθε ε, ζήτημα που θα είχε να κάνει με δικαιοδοτική εξουσία. Και άρα βρισκόμαστε σε ένα στοιχείο το οποίο περιπλέκει πιστεύω τα πράγματα. Διότι ενώ στο αστικό και το εμπορικό δίκαιο και μάλιστα ε, μέχρι και στο ε, οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο. Υπάρχουν πολύ σαφείς κανόνες ε, διάκριση των αρμοδιοτήτων και των δικαιοδοσιών μεταξύ των αρχών των διαφορών κρατών, όπου μπορεί να υπάρξει πρόβλημα από τον κίνδυνο διαφορετικής ε, ερμηνείας των τυπικών κανόνων και αυτό προκύπτει και από την σπάνια της νομολογίας του δικαστηρίου και άρα η μη προσφυγή στη δικαιοδοσία αυτή στο το πεδίο του, αστικού και του εμπορικού δικαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπεράσματα σχετικά με, τον... Ε, με την ε, ε, κυριαρχία με την έννοια δηλαδή ότι σε έναν τομέα τέτοιο που έχει λιγότερο μερίδιο από την εθνική κυριαρχία παρετούμαστε από την εθνική δικαιοδοτική αρχή εδώ έχουμε να κάνουμε στο ποινικό δίκαιο με τις εξής περιπτώσεις. Είτε πρόκειται για μια σύγκρουση δικαιοδοσιών σε περίπτωση που μια υπόθεση η ίδια μάλλον υπόθεση διαφορετικά χρονικά σημεία ε, προσάγεται σε διαφορετικά δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μπορεί να είναι αρνητική σύγκρουση, δηλαδή δεδομένου ότι δεν είναι επαρκής η κανόνες για ειδικονομική στο ποινικό αυτό ε, νομοθέτημα στον κανονισμό, γιατί δεν είναι ένας γενικός κανονισμός ε, ποινικής δικονομίας. Έχει λίγα σημαντικά αμένα, αλλά λίγα μέτρα, λίγες διατάξεις δικονομικές και άρα ε, ελήψη αυτών των λεπτομερών διατάξεων μπορεί να υπάρχει η περίπτωση για να αναφέρω εδώ τους, τις πατρίδες των ομιλούντων για να δείξω την ε, διεθνή, το διεθνικό χαρακτήρα στις υπόθεση μπορεί να έχουμε γαλλικό, ιταλικό, ισπανικό ή τι άλλο χαρακτήρα μιας δίκης με κίνδυνο ο Ιταλός ε, δικαστής να διαβάσει τον κανονισμό και να πει «Α, εγώ δεν έχω αρμοδιότητα» και μάλιστα να ε, καλέσει τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα να μεταβιβάσει τη δίκη σε ενώπιον άλλου δικαστηρίου, άλλης δικαιοδοσίας εθνικής δηλαδή, και άρα πάλι να υπάρξει αυτή η μετακίνηση τη δίκη, ώστε να μην καταλήξει ποτέ σε κανένα ποινικό δικαστήριο. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα περιθώριο χωρίς κάλυψη από δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από την άλλη θα πρέπει και ο ενδιαφερόμενος, ένας ενταλός ας πούμε υπηκός, να μπορεί είτε ε, ε, ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα να τον προσάγω σε δίκη στη Ρώμη ή το Μιλάνο και το ίδιο να είναι στο Παρίσι ή στη Μαδρίτη κόπου αλλού γιατί θα πρέπει να προσλάβει δύο δικηγόρους αλλά επίση θα βρεθεί μπλεγμένο στι συνέπειε ενό δικαιοδοτικού συστήματο, ενό ενόμου συστήματο το οποίο δεν γνωρίζει και επίση μην ξεχνάμε ότι αυτή η οδηγία PIF που δεν είναι κανονισμό και άρα δεν προσδιορίζει ε, σταθερέ ε, ποινέ, ομοιόμορφε τιμέ, θα έχει μεγάλε αποκλήσει σε σχέση με τι ελάχιστε και τι ανώτατε ε, ποινέ και άρα υπάρχει πρόβλημα λειτουργία και των. Ε, περιπτώσεων ε, της ε, ευνοϊκότερης μεταχείρισης για λόγους, ε, για ευνοϊκούς ή της, της επιβάρυνσης της θέσης του κατηγορουμένου για λόγο επιβαροντικών στοιχείων που πάλι θα εκτιμηθούν διαφορετικά σε κάθε εθνική δικαστική αρχή. Λοιπόν, το ζήτημα της επιβάρυνσης της θέσης του κατηγορουμένου δεν κρίνεται από τον δικαστή όταν αυτός θα πει «Α, εγώ θεωρώ ότι δεν με βολεύει να εφαρμόσω τον κανονισμό στο εθνικό μου δικαστήριο», αλλά σε σχέση με τον κατηγορούμενο και την επιβάρυνση της θέσεώς του ενώπιον της δικαστικής αρχής στην οποία θα προσαχθεί. Γιατί αν, λειτουργήσουμε σε ένα, αν δεν λειτουργήσουμε σε ένα σύστημα ενοπτικό, ενιαίο μετά την έγκριση του κανονισμού, αφού δεν θα υπάρχει μία ενιαία ευρωπαϊκή ποινική δικαιοδοσία θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο κατηγορούμενο να πει ότι εγώ δεν θέλω να πάω στο δικαστήριο της Μαδρίτης αλλά στο Μιλάνο. Και βέβαια αυτό μπορεί να οδηγήσει δυσκολίες. Το καταλαβαίνω. Ε, αλλά από τη σημερινή συζήτηση και ολοκληρώνω, Πρόεδρε, τι Ετέθη το ζήτημα νωρίτερα, το forum shopping, της επιλογής δικαιοδοσίας. Έχει κάποια ε, σοβαρότητα υπόθεση αυτή βεβαίω όταν προκύπτει από, τις, από τους ιδιώτες εμπλεκόμενους σε μία δίκη. Αλλά είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα εάν το forum shopping το κάνει ο εισαγγελέα. Γιατί θα βρει ότι είναι πιο ευνοϊκέ οι συνθήκε για την αποδοχή των αποδεικτικών στοιχείων, για την αξιολόγηση των επιφερειτικών ε, συνθήκων, για τη διάρκεια τη δίκη, ε, για το ένα ή το άλλο στοιχείο το οποίο επηρεάζει την εξέλιξη τη δίκη. Αυτό είναι ζήτημα τη δικαιοδοσία λοιπόν. Επίση όμω αναφέρθηκαν και πράξει που έχουν να κάνουν με την άμεση εφαρμογή του κανονισμού και σε αυτό συμφωνώ με τη Μαντάμ Blanche και κλείνω. Ε, διαδικαστικές πράξεις, διαδικαστικές πράξεις οι οποίες όχι μόνο ε, μπορούν, αλλά οφείλουν να ελεγχθούν από τον Εθνικό Δικαστή και αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μια σημαντική απόκληση από τα όσα ε, είχε σκοπό να προωθήσει το ε, σχέδιο της Επιτροπής, αλλά έχει να κάνει με την τελική διαμόρφωση της ε, διαδικασίας και των συνεπειών αυτής. Μόνο ο εθνικός δικαστής είναι σε θέση δηλαδή να αξιολογήσει τους όρους της ε, αναγνώρισης της αντικειμενικής υπόστασης ενός εγκλήματος και σε περίπτωση αμφιβολίας να ε, ζητήσει να εξεταστεί παρετέρω. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Ήσασταν και σύντομος και πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους ε, και σε όποιον θα ήθελε να κάνει ερωτήσεις προς τους προκεκλημένους μας. Δεν θέλω εγώ να τυπώσω κάποιες ερωτήσεις προς τον ε, κύριο Πατρόνα καταρχάς που μίλησε για δικαστική, ε, δικαστικό έλεγχο σε περίπτωση επικράτησης ενός μεικτού συστήματος, δηλαδή εθνικό, εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια μπορεί να έχουν συντρέχουσα δικαιοδοσία, θεωρείται ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει σε κάποιο τύπου σύγκρουση η οποία μπορεί να αποβεί εις βάρος της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εγγελίας. Και προς τον ε, Γενικό Εισαγγελέα Μπότ, θα ήθελα, μια και έγινε λόγος πάντα πάλι για την ε, δικαστική το δικαστικό έλεγχο. Τι είδους δικαστικό έλεγχο μπορούμε να έχουμε κατά τη γνώμη σας μετά όσα ακούσαμε σήμερα. Τι γνώμη έχετε εσείς. Ευχαριστώ. Α, και μετά ο κύριος Φως. Άξιλ. Ευχαριστώ. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να παρακολουθήσω όλες τις ε, τοποθετήσεις. Ελπίζω πάντως να μην σας ε, φανεί περίτη η ερώτησή μου. Να είναι ευστοχή. Καταρχάς, θέματα πιο ε, θεμελιώδη. Έχουμε το θεμελιώδη νόμο, το αντίστοιχο σύνταγμα στη Γερμανία, που ορίζει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στο φυσικό του δικαστή. Εδώ μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία σε περίπτωση ε, υπερσυνοριακών ε, αδικημάτων θα μπορούσε να επιλέξει σε ποιο δικαστήριο θα παραπέμψει τη δίκη, πώς μπορεί να τηρηθεί αυτός ο όρος του φυσικού δικαστή. Θα χρειαζόταν ένα ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο σε σχέση με τη δικαιοδοσία ή μη τι άλλο. Και η δεύτερη ερώτηση, αντίστοιχη με αυτή της κυρίας Ματέρα, πώς θα γίνεται η επαλήθευση των ε, πράξεων της Ευρωπαϊκής Εγγελίας. Υπάρχουν δικονομικοί κανόνες, ονέφερε και ο ο μιλητή μα από την Ιταλία, βεβαίω οι εθνικοί δικονομικοί κανόνε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό όργανο το οποίο πάλι κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον θα μπορούσε να αξιολογηθεί μόνο προ προς τις τη της του από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από την άλλη όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να κρίνει τις υποθέσεις. Άρα περιπλέκεται η κατάσταση, θα βρούμε άλλα νομοθετήματα διαφορετικά σε κάθε περίπτωση που θα μας οδηγήσουν στην αξιολόγηση εθνικό επίπεδο των δικονομικών διατάξεων που θα έχει τηρήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά σε περίπτωση κάποιας παράβασης ή κατάχρησης ακόμα από πλευράς της ΕΠΟ θα πρέπει να προσφύγουμε στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας έχει απασχολήσει το θέμα αυτό, έχετε κάποια γνώμη. Ναι, παρακαλώ. Βεβαίω να σα απαντήσω. Σα εξήγησα ότι είμαι υπέρ μια απόλυτα σαφούς διευκρίνησης των θεμάτων, των υποθέσεων και θα είναι ελάχιστε αυτές που θα υπαχθούν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και εκείνων των λοιπόν που βέβαια θα έχουν και τα οικονομικά ζητήματα που θα αναλαμβάνουν να κρίνουν τα εθνικά δικαστήρια. Αν λοιπόν οριστεί έτσι ο κανονισμός. Αν λοιπόν ακολουθήσει αυτή τη σαφή διάκριση, αυτή τη λύση σαφού διακρίσεω, ο κανονισμό δεν βλέπω κίνδυνο σύγκρουση δικαιοδοσιών. Τίποτε περισσότερο, εν περιπτώσει, από αυτό που βλέπουμε κατά περίπτωση είναι εδώ και εκεί αυτή την εποχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύστημα, ένα ένομο σύστημα το οποίο έχει μια τάση προς σταθερότητα και ξέρουμε βεβαίως ε, και τι, ε, σε τι παρεμβάση έχει προβεί και το δικαστήριο του Στρασβούργου. Ε, δεν θα ήθελα να επεκταθώ για να αφήσω χρόνο και για τους υπόλοιπους, αλλά Βεβαίω και στη δική μου Σύνταγμα, κύριε Φως, υπάρχει η αρχή του φυσικού δικαστή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και άρα θεωρώ ότι πρέπει να είναι σαφές εκ των προτέρων δυνάμει αυτής της αρχές του φυσικού δικαστή σε ποιο δικαστήριο θα προσαχθεί μία δίκη. Και από εκεί και πέρα ισχύουν οι εθνικές διατάξεις. Ο δόκτωρ Ράγκε, ε, εισαγγελέας ε, ε, ε Αριού της Γερμανίας, ε, μου είχε πει σε ένα συνέδριο στο οποίο συμμετάσχει εγώ, μα ξέρετε εμείς είμαστε ομοσπονδιακό κράτος και έχουμε περιπλοκές και τα λοιπά που δεν γνωρίζετε εσείς. Ε, ναι, αλλά με σαφείς διατάξεις ε, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιπλοκές. Γι' αυτό σας λέω ότι αν είναι σαφείς, σαφείς διατάξεις δεν θα προκύψουν συγκρούσεις. Παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Και πιστεύω ότι θα μπορεί να τηρηθεί η αρχή του φυσικού δικαστή. Σας ευχαριστώ, Κύριο Μπότ. Ευχαριστώ. Αν καταλάβω καλά, το ερώτημα που τέθηκε ουσιαστικά θέτει το ζήτημα της αναγνώρισης της εγκυρότητας των αποδεικτικών στοιχείων ε, που αποκτώνται σε ένα άλλο κράτος μέλος σε σχέση με την ανάθεση της αρμοδιότητας. Ε, και του που ανατίθεται η εκδίκαση υπόθεση από την εισαγγελία. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της εγκυρότητας των αποδείξεων, για μια ακόμη φορά πιστεύω ότι τα διάφορα κείμενα που υπάρχουν ε, σήμερα για τη συνεργασία, οι κανόνες και ο κανονισμός ε, θα προσθέσει κάποιες διατάξεις, άρα στην ομολογία του δικαστηρίου θα προσθεθούν διατάξεις και άλλες σε ό,τι αφορά την αρχή της αναγνώρισης. Θεωρώ ότι αυτοί οι κανόνες 99 για να μην πω 100% προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Και αν τεθούν τα προβλήματα, αυτά θα άπτονται του ενωσιακού δικαίου. Το δικαστήριο ε, πολλές φορές χρειάστηκε να καταλήξει σε αυτόνομες έννοιες. Άρα εκεί δεν ξέρω και αν πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τη δικαιοδοσία για την ερμηνεία των συνθήκων την έχει αποκλειστικά το δικαστήριο. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει και στην προκειμένη περίπτωση, στο πλαίσιο του προδικαστικού ερωτήματος. Δεν ξέρω πως και δεν κατάλαβα καλά βέβαια. τι αλλάζουμε το σύστημα. Τώρα, κάτι τελείως διαφορετικό ε, που έχει να κάνει με το νέο σύστημα είναι το κριτήριο της αστικής αρμοδιότητας, άρα του στοιχείου της εκτίμησης ε, όπου θα βασιστεί η εισαγγελία για να αποφανθεί ότι η τάδε υπόθεση που διεξαγόταν σε διάφορα κράτη θα εκδικαστεί στην τάδε δικαιοδοσία. Εκεί ίσως υπάρχουν κάποιες σκέψεις που θα έπρεπε να γίνουν και η πρώτη σκέψη ίσως είναι ουσιαστικά μια ερώτηση, να διερωτηθούμε κατά πόσον ε, η σειρά προτίμησης που επιλέγει ο κανονισμός ε, για τα κριτήρια ε, περί αρμοδιοτήτων είναι ο κατάλληλος, διότι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τελικά ότι Εκεί που έγιναν τα περισσότερα ε, περιστατικά που συνιστούν την αξιόπινη πράξη, θα πρέπει να είναι και το μέρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να ρυθμιστεί και η δικαιοδοτική αρχή. Είναι ένα κριτήριο αντικειμενικό το κριτήριο ε, του τόπου στον οποίο διαπράχθηκε το πιο βασικό αδίκημα. Είναι και ένα αντικειμενικό κριτήριο και αυτό. Και επειδή μιλάμε για απάτη, για, ε, απάτη σε βάρος των χρηματοοικονομικών σφαιρών της Ένωσης, φαντάζομαι ότι το δικαστήριο των Βρυξελών θα πρέπει να προσλάβει ε, μαζικά. Διότι μην πω ότι πρέπει να δημιουργήσει και ένα συγκεκριμένο δικαιοδοτικό όργανο που θα κρίνει, θα δικάζει τις παραβάσεις αυτές. Ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να μας προβληματίσετε περαιτέρω το όλο θέμα. Το κριτήριο της εθνικότητα του δράστη θέτει κάποια προβλήματα, ιδίως αν είναι περισσότερο του ενός. Σε πολύπλοκα δικήματα ισχύει κάτι τέτοιο. Ιδίω αυτά τα οποία θα υπόψη, τα δικήματα τα χρηματοοικονομικού τύπου. Βέβαια, έχουμε και μια υπόθεση που πρέπει να προσθέσουμε ότι ο δράστης θα μπορούσε να είναι και υπήκοστερο του κράτου. Τότε τι κάνουμε. Πρέπει να υιοθετήσουμε κάποιο άλλο κριτήριο. Η κατοικία, το διαμονή διαμονής του δράστη. Γιατί αυτού θύματο όμω. Τι να πω. Καλή τύχη πάλι για το δικαστήριο των Βρυξελών. Όπως καταλαβαίνετε, μη δύο, αλλά ε, νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε με τον Ιταλό συνάδελφο. Σίγουρα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε και το εξής. Πρέπει να δούμε και το γενικό θέμα της συνεργασίας, της δικαστικής συνεργασίας που τίθεται αλλά οι δικαστές που μελετούν και εκδικάζουν αυτές τις υποθέσεις και οι εισαγγελείς δεν είναι πια και κακόπιστοι όλοι. Δεν ξυπνάνε κάθε πρωί και σκέφτονται πόσα θεμελιώδη δικαιώματα σήμερα θα παραβιάσω. Έτσι δεν είναι. Και ξανά μη δυο. Διότι είναι σαφές ότι συμμετέχοντας πλήρως στη δικαστική, στην εθνική αλληλέγγυα δικαστική δράση Εδώ μιλάμε κυρίως για το σεβασμό του κράτους δικαίου και αυτό ε, κινεί τους ε, δικαστές. Πρέπει να γίνονται σεβαστές αρχές του κράτους δικαίου, τόσο ε, εσωτερικό έλεγχο. δεν απέναντι τεταμένο σε να βάλτε το αλλού αυτό. τι θα κάνει το μόνιμο σώμα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τελικά όλοι θα, θα είναι συνένοχοι τελικά σε αυτή την καταπάτηση των αρχών του κράτους δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι για μια ακόμη φορά έχουμε το σύστημα της συνθήκης, την εθνική δικαιοδοσία, με τις εγγύσεις της. Και αν τι να πω, αν συμβεί κάτι σε μια χώρα, τι να πω, είναι μέρος της Ένωσης, υπάρχουν βάσεις, κοινέ. Πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές του κράτους δικαίου. Οι αναπαλωτρίωτες αρχές του κράτους δικαίου. Αλλιώς δεν μπορεί να ενταχθεί κάποια χώρα σε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω, μήπως μου ξέφυγε κάτι. Μπα, δεν φαντάζομαι. Πρέπει να το δεχθούμε λοιπόν. Και ολοκληρώνω. Αλλά δεν μπορώ να μην πω και κάτι για αυτήν την ιδέα. Πριν την έναρξη δίωξη να υπάρχει ξεχωριστό έλεγχο από το δικαστήριο. Τι να πω, όλα είναι ε, πιθανά ε, υπό τον ήλιον. Ε, τα πάντα μπορεί να φανταστεί κανεί. Αλλά αυτόν τον έλεγχο πότε θα τον κάνει το δικαστήριο. Όταν θα πει εισαγγελία η Ευρωπαϊκή, εγώ αποφασίζω να προχωρήσω σε δίωξη. Και πού υποβάλλεται, πού δημοσιεύεται, ποιος ε, πού θα μπορούν οι διαφερόμενοι να ε, υποβάλουν τις ενστάσεις τους ενδεχομένως. Άρα δεν προχωρούμε σε δίωξη και τελειώνουμε. Έχουμε μια καταγγελία για παράδειγμα. Από την Όλαφ. Καταγγέλει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ο τάδε Δίνα ή το τάδε σύστημα δεν φαίνεται καθόλου καθαρό το πράγμα. Πρέπει να το ερευνήσετε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεδριάζει ε, υπό το, μόνιμο σώμα, δεν ξέρω εγώ, ε, μαζικά συλλογικό συλλογικό όργανο και λέει, αποφασίζει ότι φαίνεται η τάδε δίνα εταιρεία να έχει διαπράξει απάτη στο ό,τι αφορά τον κοινοτικό ΦΠΑ και σε σημαντικό βάθμο. Πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της δίωξης. Ποιος θα ενημερώσει τους θυγόμενους. Σε ό,τι αφορά τον προτέρων έλεγχο των ε, διώξεων, ποιος θα πει ότι σας κοινοποιώ ότι θα σας ε, διώξουμε στο πλαίσιο μπλα μπλα μπλα, ε, γιατί στην τάδε χώρα. Επιλέγω γιατί αυτή η χώρα, ε, γιατί αυτή είναι η δικαιοδοσία. Άρα καταργείται κάθε έννοια, δεν γίνεται καμία δίωξη, τέρμα, σταματάνε οι εργασίες. Γιατί δεν πρέπει να γίνει καμία έρευνα ποτέ υπό τέτοιε συνθήκε, αν κάτι δημοσιοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Που μπορεί θεωρητικά άρα όλα αυτά που λέμε να είναι πολύ έτσι ωραία και καλά, αλλά στην πράξη αντιπαραγωγικά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους δεκεκριμένους ομιλητές μας. Παρακαλώ τον Άξελ Φως, τον συνάδελφο μας με τον οποίο πριν από μερικούς μήνες αποφάσισαμε να οργανώσουμε αυτό το, το, αυτή την ακρόαση. Αν θέλεις να έρθεις εδώ, έχουμε μια θεσούλα εδώ στην άκρη, αν θέλεις να έρθεις εδώ. Ένα αναμονή της Επιτρόπου Γιώργου αρμόδιας για θέματα δικαιοσύνης, ισότητας των φίλων. Άξελ. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Ε, από όσο βλέπω εγώ. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως αποκομίσαμε σήμερα την ε, κατεύθυνση που θα πρέπει να λάβει εν τέλει η οδηγία ΠΙΦ, την ανάγκη για σαφής κανόνες για τις δικαιοδοσίες, όλα αυτά για να υπάρξει μια αποτελεσματική ε, διαρρύθμιση χωρίς πολλά προβλήματα του τρόπου λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικά εν τέλει. τα όργανα και βέβαια τα όργανα αυτά θα έχουν το καθένα τις δικές του αρμοδιότητες μένα, αλλά θα χρειαστεί και ένα βαθμό ευελιξίας. Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα της κατανομής των δικαιοδοσιών μεταξύ των όσων προβλέπει η ΠΙΦ προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ΕΠΟ, την Eurojust, Όλαφ, εθνικές αρχές με διαφορετικά επίπεδα αρμοδιοτήτων για την κάθε μία και άρα εκεί θα χρειαστούν κανόνες αφής ώστε να μην πέσει σε αντιφάσει στο σύστημα, να μην φέρει τον έναν απέναντι στον άλλον τη δικαιοδοσίε και να μην δυσκολέψει την ε, αποτελεσματικότητα του έργου τους. Για την Όλαφ ίσως χρειάζεται να μας απασχολήσει πιο προσεκτικά αυτή η υπόθεση, γιατί δεν έχει μόνο αυτά τα καθήκοντα η Όλαφ και άρα ίσως θα μπορούσαμε σε ένα εσωτερικό διάλογο να βρούμε κάποιες άλλες λύσεις. Η Όλαφ μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης, μπορεί να αποτελέσει ένα ε, συμβουλευτικό όργανο για την ε, ΕΠΟ με την υποστήριξη την επιμελητιακή ακόμη ακόμη, αλλά βέβαια και στη Eurojust μπορεί να στραφεί η ΕΠΟ για, την, ε, για τα οργανωτικά της οργανωτικές ανάγκες. Πρέπει να τα κοιτάξουμε εις βάθος και να δούμε πώς αυτές οι διαφορετικές ε, δομές μπορούν να αναπτυχθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό. Θα υπάρχει και ένας ε, μηχανισμός συντονισμού και νομίζω αυτά λίγο πολύ από πλευράς μου. ως πρόταση για να προχωρήσουμε προς ένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Φως. Και καλώς ορίζω την Επίτροπο Βέρα Γιώροβα, Επίτροπο για Δικαιοσύνη και Ισότητα των Φίλων. Σε ευχαριστώ που έρχεστε να λάβετε μέρος στις εργασίες μας, οι οποίες βέβαια καταλήγουν σε λίγο, αλλά είναι πολύ σημαντική και πολύτιμη για όλους μας η δική σας τοποθέτηση. Σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Στο κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη που ήρθα αργά, διότι βλέπετε μόλις επέστρεψα από Λισαβόνα. Καθυστέρησε η πτήση μου λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν στις Βρυξέλλες. Πριν φύγει το αεροπλάνο για να έρθει να μας πάρει. Και μετά στην επιστροφή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τη δυνατότητα που δίνετε να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση ο χρονισμός είναι έξοχος, διότι τώρα φτάνουμε στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα το Κοινοβούλιο θα πρέπει σύντομα να δώσει τη συνένεσή του. Και θυμάμαι ακόμα τις πρόσφατες συναντήσεις που είχαμε στους Πορτογάλους συναδέλφους, τις ζητήσεις που είχαμε. Η επίσκεψή μου στην Πορτογαλία εστιαζόταν πολύ σε αυτό το θέμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Έχει επιτευχθεί καλή πρόοδος από το Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη εξέφρασαν την στήριξή τους καταρχήν για διάφορα βασικά συστήματα του προτινόμενου κανονισμού και φαίνεται ότι είναι καθοδόν προς ε, το να καταλήξουν σε γενική προσέγγιση του έτους. Βασίζομαι στην επικείμενη Σλοβακική Προεδρία να είναι ένα ισχυρό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια. Ήδη συζήτησα με τον Σλοβάκο Υπουργό, τον νέο Υπουργό της νέας κυβέρνησης, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι έτοιμος να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο από την Ολλανδική Προεδρία, την οποία πρέπει να ευχαριστήσω. Οι συνάδελφοι από την Ολλανδία πραγματικά σημειώσαν σημαντική πρόοδο. Στόχος όσον αφορά το περίπλοκο θέμα της δύσκολης διαπραγματεύσης ήταν και παραμένει να έχουμε έναν ανεξάρτητο φορέα, ανεξάρτητη και δυνατή εισαγγελία. Θα πρέπει να προστατεύει καλύτερα τα οικονομικά συμφέροντά μας σε όλη την Ένωση. Πρέπει να δώσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τους εμπλεκόμενους φορείς, για τους φορολογούμενους, για όλους. Και συζητήσεις με τους υπουργούς και τους γενικούς εισαγγελείς και τους εμπειρογνώμονες πάντα τόνιζα ένα κρίσιμο θέμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αντικαθιστά τις, ευρω... τις εθνικές εισαγγελίες. Πρέπει να οικοδομηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο, σαν, ένα... σαν μια πρόσθετη στιβάδα αρμοδιοτήτων, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν εύκολα σε εθνικό επίπεδο εθνικέ εισαγγελίε, γιατί μιλάμε για μεγάλα εγκλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα πολύ συχνά. Για να πετύχουμε λοιπόν τον στόχο της δημιουργίας ισχυρής και ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα φέτος. Πρώτα απ' όλα οι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητες, ξεκάθαρες. Πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση των αρμοδιοτήτων. Χρειάζεται ισορρόπηση, εξισορρόπηση των αρμοδιοτήτων να, μην, ε, να έχει τελικά αρμοδιότητα και υποθέσει ΠΙΦ και δεν θα πρέπει να έχουμε περίπλοκο καθεστώς ούτω ώστε να είμαστε αναποτελεσματικοί και να γίνονται παράλληλε μακροσκελείς έρευνε. Τέλος Ιουνίου θα γίνει μια συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες από αρκετά κράτη-μέλη. Θα είναι έλεγχος πραγματικότητας όπως το αποκαλούμε. Θέλουμε να δούμε ποιε είναι οι αρμοδότητες, ποια είναι η δομή, ποιο είναι το μοντέλο του EPPO, ω έχει τώρα. Θα δούμε λοιπόν την ε, οργανωτικά θέματα, οικονομικά θέματα, θέματα προσωπικού και θα κάνουμε τον έλεγχο της πραγματικότητας, θα αποτιμήσουμε το όλο εγχείρημα. Θα πάρουμε μια υπόθεση και θα την δοκιμαστικά, θα κάνουμε προσημείωση αν θέλετε, θα την περάσουμε μέσω του μηχανισμού του EPPO και θα δούμε πού βρισκόμαστε. Θα δοκιμάσουμε το μοντέλο του ΣΥΠΗΝ, να δούμε το μοντέλο που προτείνουμε είναι εύρυθμο. Και προτείνω να διοργανωθεί αυτός ο έλεγχος πραγματικότητας, ούτω ώστε να γίνει κάπου σε μια ευρωπαϊκή φυλακή, για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι κάτι που θα έχει να αντιμετωπίσει ανθρώπους, ανθρώπινα όντα, ανθρώπους που κατηγορούνται για ποινικά δικήματα. Να καταλάβουμε ότι η διαδικασία δεν θα πρέπει να είναι πολύ περίπλοκη ούτε μακροχρόνια, διότι είναι συμφέρον μας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποδίδει δικαιοσύνη εγκαίρως. Δεύτερον, και είναι κάτι που γνωρίζω από τις συζητήσεις με την εισηγήτρια την κυρία Ματέρα και μερικούς από εσά, θέλω να επιβεβαιώσω σήμερα ότι είμαστε πεπισμένοι ότι το ΦΠΑ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο της οδηγίας ΠΙΦ και άλλε αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έχουμε σαφή επιχειρηματολογία που έχει επιβεβαιωθεί και από το ΔΕΚ και θα πρέπει να το ακολουθήσουμε. Τρίτον, θα πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου τις λεπτομέρειες της δομής, ανησυχούμε όσον αφορά τα αποτελέσματα της εθνικοποίησης, αν θέλετε, τι γίνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων που είναι σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η αρχή, της, η αρχή του εθνικού συνδέσμου, αν παραμείνει αυτή η αρχή, θα πρέπει να δίνει δυνατότητα τουλάχιστον να επανανατίθενται ε, υποθέσεις αν είναι να λειτουργεί εύρυθμα η υπηρεσία, κυρίως αν υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας υποστηρίζω τη δημιουργία μονίμων δικαστηρίων, αλλά πιστεύω ότι η αρμοδιότητά τους ίσως να μειωθεί μέσω της εισαγωγής της δυνατότητας ανάθεσης των αποφάσεων σε διάφορους Ευρωπαίους εισαγγελείς για υποθέσεις κάτω από 100.000 ευρώ. Μια τέτοια ανάθεση εξουσιών υπονομεύει τον φορέα που δημιουργούμε. Θα πρέπει αυτό να αφορά ίσονες περιπτώσεις ούτως ώστε να, το κεντρικό επίπεδο να μπορεί να υποπτεύει και να έχουμε μια πραγματική πολιτική δίωξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέταρτον, θέλουμε να έχουμε να διαφυλάσσουμε τα διδικαστικά δικαιώματα των διοκόμενων και των κατηγορουμένων, δικαίωμα νομικής αρρωγής το δικαίωμα να παρουσιάσουν αποδείξεις και να ζητήσουν από την εισαγγελία να συλλέξει αποδείξεις, κάτι πρώτην αρχικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά θα πρέπει να επιστρέψουν στον κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση και τις εξουσίες της αγγελίας. Οι διαδικαστικές ρήτρες διαφύλαξης θα πρέπει να προβλέπουν πρόσθετες εγγυήσεις που θα αντισταθμίζουν τις ευρωπαϊκές εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, τα δικαιώματα των υπόπτων και των διαφόρων ατόμων σύμφωνα με εθνικό νόμο που εναρμονίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες δεν είναι κάτι υπαρκή εδώ. Πέμπτον, βλέπω να υπάρχει σαφή σχέση μεταξύ της προστιθέμενης αξίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της αρμοδιότητας να καλύπτει και τις υποθέσεις απάτης ΦΠΑ. Το νομικό πλαίσιο είναι σαφέστατο, κυρίως μετά ε, τις διάφορες αποφάσεις. Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι οι διασυνοριακές υποθέσεις ΦΠΑ κάποιες διάστασεις θα πρέπει να καλύπτονται. Και αυτό είναι το θέμα των συζητήσεων με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης. Ήδη συζήτησα με κάποιους Υπουργούς Οικονομικών γι' αυτό, διότι θα πρέπει να κατανοήσουν το ότι αυτό που ετοιμάζουμε ποιοι είναι. Πολλοί υπουργοί οικονομικών πιστεύουν ότι αυτό είναι θέμα φόρου, φορολόγησης. Και αυτό είναι καθήκον μου. Και καθήκον στου συναδέλφου θα κάτι μέσα εξηγήσουν θέμα ποινική δικαιοσύνη, αυτό που εξετάζουμε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Πρέπει να κατανοήσουμε τη διάσταση αυτή. Συζητήσαμε με του υπουργού και του γενικού εισαγγελεί το πεδίο εφαρμογής και τον χαρακτήρα της απάτης ΦΠΑ που θα πρέπει να ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία και η θέση μου είναι σαφής. Η διασυνοριακή απάτη μεγαλύτερης κλίμακας όπου οι εθνικές αρμοδιότητες και οι εθνικοί φορείς δεν μπορούν να ερευνήσουν και να διώξουν αποτελεσματικά κάτι που ξεπερνά τις εξουσίες τους και τις δυνατότητές τους και τους περιφερειακούς τους περιορισμούς είναι αυτό. Βλέπω σαφώς λοιπόν ότι αυτό που μου λένε οι υπουργοί είναι ότι για τέτοιες περιπτώσεις δημιουργούν κοινέ ερευνητικές ομάδες. Αυτή είναι η παρούσα μέθοδος που χρησιμοποιούν για διασυνοριακή διερεύνηση απατών και εγκλήματος ΦΠΑ και συμφωνούν μαζί μου όταν τους λέω ότι αυτές οι μικτές ερευνητικές ομάδες δημιουργούνται κατά περίπτωση για κάθε υπόθεση. Εάν έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα έχουμε μια ευρωπαϊκή ισχυρή ομάδα που θα ερευνά αυτές τις απάτες, αυτά τα εγκλήματα και αυτή η ομάδα θα έχει θεσμική μνήμη και συνέχεια και αυτό δίνει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή ιδιαίτερη δυναμική. Είμαι πεπισμένη ότι θα είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα και ίσως και φθηνότερα και σίγουρα αποτελεσματικότερα ε, αποτελεσματικότερο εργαλείο να χρησιμοποιηθεί για τη διασυνοριακή απάτη όσον αφορά το ΦΠΑ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ε, ζητήσω την διακομματική σας υποστήριξη για όλα αυτά τα θέματα. Όπως σας είπα, είναι περίπλοκο το χαρτοφυλάκιο. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και από διάφορους τομείς, δικαιοσύνη ή το τομέα των οικονομικών. Ελπίζω ότι μπορούμε να, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον αφορά τον κανονισμό για το Eurojust, ούτως ώστε να επικαιροποιήσουμε και να βελτιώσουμε την λειτουργία αυτού. Είναι και η ώρα να προχωρήσουμε όσον αφορά το Eurojust. Οι διαπραγματεύσεις για το θέμα του EPPO, της Ευρωπαϊκής Εγγελίας, φτάσαν σε μια φάση όπου οι σχέσεις μεταξύ του Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εγγελικής Αρχής φαίνονται σαφέστερα, πιο ξεκάθαρα και θα πρέπει να καταλήξουν σε μια συμφωνία όσον αφορά τον κανονισμό μέχρι το τέλος ενεστώτος έτους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε πολύτιμη παρέμβασή σας, ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Πάντα καταφέρουμε να συνεργαζόμαστε από αυτών των ζητημάτων και όχι μόνο από αυτών. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος αυτής της διασκέψεως, αυτής της ακροάσεως. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη συμμετοχή σας σαν εισηγήτρια ε, για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής μαζί με τον συνάδελφο Axel Vox για τη μεταρρύθμιση του Eurojust στο Ευρωκοινοβούλιο Θέλουμε να νικήσουμε αυτή την πρόκληση στο πεδίο της δικαστικής συνεργασίας σε θέματα ποινικά. Θέλουμε να έχουμε ε, μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή που θα είναι ισχυρή, αποτελεσματική και μεταρρύθμιση του Eurojust με ένα Eurojust που θα μπορεί να γίνει ισχυρότερο μέσω μιας νομικής βάσης και μέσω πολύ μεγαλύτερων πόρων. Εν γέννη, οι προκλήσεις που καθορίζουμε είναι κάτι που προσπαθούμε πάντα να τις πετυχαίνουμε και μετά να προτείνουμε νέες προκλήσεις. Λοιπόν, θα ενημερωθούμε τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ όλους τους επιφανείς ομιλητές που συμμετείχαν σε αυτή την ημερίδα εμβάθυνσης και ανταλλαγής απόψεων και συστάσεων και ενημέρωσης που ήταν πάρα πολύ πολύτιμο όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.